Dear colleagues, good morning. Uh, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. We'll continue the work. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το κύριο θέμα μας σήμερα είναι η δημόσια κρόαση για την πολιτική συνοχής και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Μάλιστα θα συντάξουμε και έκθεση πρωτοβουλίας με το θέμα αυτό. Η κυρία Ρέντκε είναι η συγγήτρια. Θα πρότεινα λοιπόν να συζητήσουμε από κοινού αυτά τα δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης, την έκθεση Ρέντκε και τη δημόσια κρόαση. Η νομοθεσία για την πολιτική συνοχή προβλέπει χρηματοοικονομική υποστήριξη για ε, άπορες κοινότητες ε, στις, ε, στην Ήπεθρο και στις αστικές ε, ζώνες γιατί το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εδαφική προσέγγιση ε, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 προβλέπει νέες δυνατότητες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων και στόχων που θα προωθούν τη θέση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και θα έχουν τοπικό προσανατολισμό. Έχουμε μοιράσει ξεχωριστά το πρόγραμμα της δημόσιας ακρόασης. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους καλεσμένους μας για ένα δεκάλεπτο στον καθένα. Και κατόπιν θα καλέσω την εισηγητριά μας, την κυρία Ρέτκε, να μας κάνει την παρουσίαση της ε, έκθεσής της. Θα ακολουθήσει γύρω συζήτησης ε, με σχόλια και ερωτήσεις από τους συναδέλφους και στο τέλος θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια Ρέντκε για τα συμπεράσματα. Η διορία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση Ρέντκε είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2015 στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου. Αν ε, ληφθούν εμπρόθεσμα, αν υποβληθούν εμπρόθεσμα οι τροπολογίες, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου. Επίσης, μετά το πέρας ε, της πρωινή μας συνεδρίασης και γύρω στις 12.30 η κυρία Ρέντκε θα, θα ε, οργανώσει μια μικρή δεξίωση ε, έξω ακριβώ από την αίθουσα της συνεδρίασης. Αυτό το κοκτέιλ θα παραθέσει η κυρία Ρέντκε κατά τις 12.30 αμέσως έξω από την αίθουσα. Για να μην χρονοτριβούμε, όλο θα δώσω πρώτα το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Άννα Κράστεβα, που είναι η Διευθύντρια του ΣΕΡΜΕΣ, του Κέντρου για τους Πρόσφυγες, τη Μετανάστευση και τις ε, Εθνικές σπουδέ στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο. Έχετε το λόγο κυρία Κράστεβα για 10 λεπτά. Είναι σχεδόν αδύνατο να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε μέσα σε 10 λεπτά το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Εγώ θα, θα περιοριστώ γύρω σε τρία θέματα, θα περιστραφώ γύρω από τρία θέματα. Το γιατί, το ποιος και το πώς. Καταρχήν, η τροτότητα, η ευπάθεια των πληθυσμών δεν σχετίζεται μόνο με την ασφάλεια, ανασφάλεια ή τη φτώχεια, αλλά και τον κίνδυνο και την αξιοπρέπεια. Και αυτό το θέμα βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών και αποτελεί και πολύ επίκαιρο και μείζωνα πολιτική πρόκληση. Γιατί η βασική μου θέση ε, προβλέπει ότι το πρόβλημα των Ρωμά δημιουργήθηκε για πολλούς ε, διάφορους και περίπλοκους λόγους. Από όλο αυτό το πλέγμα των λόγων θα σταθώ σε δύο. Τους πολιτικούς ε, και τους πολιτιστικούς πολιτικούς, όχι από ανθρωπολογική άποψη, αλλά από πολιτική κουλτούρα άποψη. Η τροτότητα, η των Ρωμά είναι ένας εκλογικό πόρος ουσιαστικά για τις πολιτικές ελίτ. Μπορεί να σας σοκάρει αυτή η διαπίστωση, αλλά θα αναπτύξω την ιδέα μου γιατί έχει πολλές πτυχές. Καταρχήν συμβολική πτυχή, γιατί η ρητορική κατά τον Ρωμά κινητοποιεί κυρίως ακραίες εξτρεμιστικές ακροδεξιές ε, οργανώσεις και κόμματα. Η τροτότητα όμως των Ρωμά ε, έχει και μια κυριολεκτική έννοια. Και έχουμε πολλά μετακομμουνιστικά κόμματα σε πολλές χώρες ε, που προσπαθούν να προσελκύσουν την ψήφο των Ρωμά. Και το τονίζω αυτό γιατί όταν λέμε πολιτική συνοχής ε, σκεφτόμαστε κυρίως τη δημόσια διάσταση αυτής της πολιτικής. Έχουμε όμως κυρίως ε, την πολιτική ιδεολογία περισσότερο και το πώς οι πολιτικοί ε, και όχι οι πολιτικές υποφελούνται από την τροτότητα, τον ευάλωτο χαρακτήρα των κοινοτήτων Ρωμά. Ο δεύτερος λόγος είναι πιο θεωρητικός, αλλά οι πολιτικές έχουν αλλάξει αισθητά. Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η έννοια του άλλου είχε πολιτική, ιδεολογική διάσταση, αλλά στην ε, περίοδο μετά τον ψυχρό έχουμε τον άλλο ε, να προσδιορίζεται περισσότερο από εθνοτικές, ε, πολιτιστικές, θρησκευτικές συνιστώσεις. Και έτσι αυτή η ρητορική κατά το Ρωμά και η συμπεριφορά λαμβάνει άλλη τρόπη. Για όλους αυτούς τους λόγους οι Ρωμά έχουν ε, γίνει all exclusive από κάθε άποψη δηλαδή, από οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και συμβολική. Είναι απόκληροι ουσιαστικά οι Ρώμα, αποκλείονται από παντού. Έχουμε βέβαια και τους πρόσφυγες, τους νέους Ρωμά όπως τους αποκαλώ, που επίσης είναι αποκλεισμένοι και τη χανούση μεταχείριση στην πολιτική ρητορική, παρόμοια με τους Ρωμά δηλαδή, είναι και αυτοί αποκλεισμένοι, περιθωριοποιημένοι. Και στις συζητήσεις ε, και οι πρόσφυγες και οι Ρωμά ε, θεωρούνται υπό την προοπτική του γκέτο, των καταβλισμών υπό την έννοια του homo sacer, του agamben, του ανθρώπου δηλαδή που είναι ταυτόχρονα ιερός και καταραμένος. Ποιοι είναι τώρα οι βασικοί φορείς, ποιοι είναι ε, οι κύριοι πέτοι αυτής της ε, τροτότητας των Ρωμά. Η βασική πέτοι είναι η πολιτική. Αυτή είναι κυρίως υπεύθυνη για τον ε, ευάλωτο χαρακτήρα των Ρωμά. Και εδώ δίνω δύο παραδείγματα. Αναφέρω μια χώρα, θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο παντού. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε για τελείως ασήμαντους λόγους, για δυνατή μουσική, για θόρυβο. Ξεκίνησε μια σύγκρουση που απέκτησε μεγάλες διαστάσεις και δημιούργησε μία ένταση της κατάστασης και της πολιτικής και της κοινωνικής στην χώρα αυτή. Στην ίδια χώρα, σε μία άλλη πόλη που έχει παρόμοια δημογραφική και οικονομική σύσταση, έχουμε μία γειτονιά Ρωμά, όπου οι Ρωμά στεγάζονται σε κανονικές κατοικίες, σε κανονικά σπίτια, οι γονείς εργάζονται και μάλιστα έχουν και μία αργία, μία γιορτή που αποδίδουν και βραβείο του έντιμου Ρωμά σε δημόσιες προσωπικότητες της κοινότητας Ρωμά. Ο δεύτερος φόρος, ο δεύτερος παράγοντας, μπορεί να ακούγεται παράδοξος και θα το τονίσω αυτό πιο, για την υπευθυνότητα ε, της τροτότητας αυτής. Η νεολαία είναι ο πιο ενθουσιώδης ε, φορέας αυτής της κινητοποίησης κατά της φτώχειας. Αν όμως θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η κινητοποίηση, κατά της φτώχειας συνιστούν ένα πολύ μικρό τμήμα της κινητοποίησης της νεολαίας γενικώ. Η σύγχρονη νεολαία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες περισσότερο ασχολείται με τα βουνά, με, τα, με την προστασία των πτηνών, με οικολογικά θέματα, με οικολογικό προβληματισμό. Περισσότερο για τέτοια θέματα, οικολογικά και περιβάλλοντος κινητοποιείται παρά κατά τις φτώχειας. Άλλο παράδοξο, το ίντερνετ. Το ίντερνετ βέβαια δεν είναι παράγον, είναι ένας χώρος, αλλά θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερος τον τεράστιο ρόλο του ίντερνετ ε, σε ό,τι αφορά τη διόγκωση της ξενοφοβίας. Η ξενοφοβία στο δημόσιο χώρο ε, ε, ε προωθείται περισσότερο μέσω του ίντερνετ. Γιατί πριν από το ίντερνετ δεν υπήρχε τόσο μεγάλος χώρος που μπορούσε να, προβληθεί, να προβληθούν αυτές οι ξενοφοβικές δυνάμεις. Και επίσης έχουμε και τις ελίτ των κοινοτήτων Ρωμά, που είναι βασικός παράγοντος που διαρωτόμαστε είναι έτοιμα της λύσης ή έτοιμα του προβλήματος τελικά, η ελίτ Ρωμά. Τώρα, με ποιο τρόπο. Κάθε δημόσια πολιτική ξεκινά με το βασικό ερώτημα ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της και της πολιτικής συνοχής για το θέμα των Ρωμά. Οι πρώτες τρεις είναι ουσιαστικά η εξής μία, η παιδεία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει μια κοινωνία της γνώσης. Πώς όμως μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία της γνώσης με αναλφάβητους εργαζόμενους. Mm. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το παράδοξο. Γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον 20ο αιώνα προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τον αναλφαβητισμό, αλλά ο 21ος αιώνας έχει δημιουργήσει ένα νέο αναλφαβητισμό. Είναι αδύνατο να ξεπερασουμε τον αναλφαβητισμο αλλα ο 21 ο αιωνας εχει δημιουργησει ενα νεο αναλφαβητισμο ειναι αδυνατο να δημιουργήσουμε μια κοινωνία της γνώσης με αγράμματους, αναλφάβητους εργαζόμενους. Οπότε μπορούμε να έχουμε νέες φιλοδοξίες ε, της δημόσιας πολιτικής χωρίς να να έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος ή από τα μαθήματα του παρελθόντος. Γιατί είχαμε μια δεκαετία φιλόδοξων πολιτικών που ολοκληρώνονται φέτος και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Γιατί και η Παγκόσμια Τράπεζα και διάφορα θεσμικά όργανα ε, δημοσίασαν ε, ε, μελέτες τεκμηριωμένες που δείχνουν παρά τη δεκαετία αυτή φιλόδοξη πολιτική διάκριση εις βάρος των Ρωμά. Αυτά τα συμπεράσματα τα γνωρίζαμε φυσικά ούτως ή άλλως και πριν τις μελέτες. Αυξάνεται η φτώχεια, αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, ε, η έλλειψη ενοχής μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και αν δεν διδαχθούμε από τα παθήματα του παρελθόντος και από τα λάθη μας και τις αποτυχίες μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τοπικές αρχές. Ήδη αναφέρθηκα σε δύο είδη εμπειριών και μερικές φορές είναι ο ίδιος ο δήμαρχος που κάποια στιγμή εφαρμόζει την πολιτική της κοινωνικής ένταξης με αξιέπαινες πρακτικές για την εκπαίδευση, για την απασχόληση και ταυτόχρονα ο ίδιος κάποια άλλη στιγμή, ο ίδιος Δήμος στην ίδια πόλη, ο ίδιος Δήμαρχος στην ίδια πόλη, εφαρμόζει πολιτικό αποκλεισμό, οργανώνοντας για παράδειγμα ένα δημοψήφισμα που αποκλείει τους ψηφοφόρους Ρωμά. Οπότε μια πολιτική θα πρέπει να δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να μην αφιταλαντεύεται ο ίδιος ο Δήμαρχος μεταξύ ένταξης και αποκλεισμού, αλλά να διαλέγει πάντα το ίδιο θέμα, την ένταξη. Και έχουμε και κάποιες καλές πρακτικές. Να σταθώ σε μία που την αποκαλώ all inclusive, όλα μέσα, όλοι στην ένταξη. Είναι μία πρακτική μικρής εμβέλειας, αλλά εμπλέκει όλα τα βασικά θέματα και τους βασικούς παράγοντες. Πρόκειται για την πολιτική της υγείας, που είναι από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής. Ε, η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται από την κοινωνία των πολιτών στα περισσότερα στοιχεία από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και από πανεπιστημιακούς κύκλους, από τα πανεπιστήμια. Επίσης, να δημιουργείται ένα πολυφωνικό, ε, πολυσχηδές αποτέλεσμα και για τους Ρωμά, δηλαδή να μορφώνονται, να σπουδάζουν οι Ρωμά και να γίνονται γέφυρες μεταξύ της δικής τους κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Να γίνονται υποδείγματα, δηλαδή μοντέλα, πρότυπα, είναι πολύ θετικό ένα τέτοιο μήνυμα και αποδεικνύει ότι υπάρχουν τελικά καλές πρακτικές. Επίσης, γιατί η κοινωνία των πολιτών δεν είναι πιο καινοτόμα. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα πιο καινοτόμα, πιο αποτελεσματική. Και ακόμη και μερικές φορές και από τους νομοθέτες, από τους ηθήνοντες των πολιτικών. Να σας υπενθυμίσω το χρόνο μόνο, κοιτάτε και λίγο το ρολόι σύντομα να ολοκληρώσω. Ένα πολύ καλό παράδειγμα που δείχνει άλλο ένα επιτυχημένο μείγμα ε, εθελοντισμού, ε, δημιουργικότητας, τέχνης, πειραματισμού. Και μία σημαντική αλλαγή που πρέπει να έρθει με το πρασίνισμα κατά κάποιο τρόπο της κατά των διακρίσεων. Θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστική αυτή η κινητοποίηση, όπως είναι και η περιβαλλοντική οικολογική. Και στο διαδίκτυο και εκτός. Και επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο για την κινητικότητα των Ρωμά, τη μετακίνηση των Ρωμά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρείται ως σημαντική πρόκληση, μίζωνα πρόκληση, και πρόβλημα για πολλές πόλεις. Αν το δούμε όμως αυτό υπό τη σκοπιά των Ρωμά, πολύ συχνά είναι και θα μπορούσε να είναι σημαντικός πόρος για χειραφέτηση, για ανέβρεση εργασίας, για δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα παιδιά θα μπορούν να σπουδάζουν, να πηγαίνουν στο σχολείο και που οι γονείς θα απασχολούνται όχι στην παραοικονομία, αλλά σε επίσημες θέσεις απασχόλησης, ώστε να δημιουργηθεί πραγματική κοινωνική ένταξη. Και ποια είναι εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση μιας επιτυχημένης πολιτικής. Φυσικά δεν θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθούν από τη σελίτη Ρωμά, αλλά να γίνουν πιο υπεύθυνε οι ελίτ απέναντι στους Ρωμά. Και αυτό θα πρέπει να πούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η ένταξη των Ρωμά εξαρτάται πρώτα απ' όλα από, ισχυρή, από την ισχυρή πολιτική θέληση. Δεν μπορούμε με το ένα χέρι να δίνουμε πολιτική συνοχή και από το άλλο να έχουμε στρατηγική εις βάρος των Ρωμά. Θέλουμε ισχυρή πολιτική βούληση για να ξεπεράσουμε τον αποκλεισμό. Οπότε η πολιτική συνοχή θα είναι επιτυχής και αποτελεσματική μόνο αν συνδυαστεί με καινοτόμες πρωτοβουλίες κοινωνίας των πολιτών και να ολοκληρώσω με κάτι που είπε ένας από τους μεσολαβητές της υγείας όταν έλαβε το πολιτήριο, είπε ότι δεν μπορεί κανείς να διαλέξει τους γονείς του και πού θα γεννηθεί, αλλά μπορεί να διαλέξει τι θα γίνει στη ζωή του χρειάζεται μια αποτελεσματική πολιτική και ίσως και ένα τάτς ουτοπίας που να μας επιτρέψει να πιστεύουμε ότι η επιτυχία είναι δυνατή. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Και τώρα με ιδιαίτερη χαρά να δώσω το λόγο στην κυρία Καρολίνα Φερνάντες, που είναι αναπληρώτρια διευθύντρια ε, του Ιδρύματος Σεκρεταριάδο Χιτάνο, Γραμματέία των Αθηγάνων και Ρώμα. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που σήμερα στην Επιτροπή και να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σύνταξης αυτής της έκθεσης καθώς και την ευκαιρία που μας δίνεται να παρακολουθήσουμε την... Ε, να παρακολουθήσουμε την έκθεση από την αρχή της σύνταξής της και που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω τη γλώσσα μου θα μιλήσω στα ισπανικά. Θα σας παρουσιάσω αυτή την υπόθεση από την άποψη της εμπειρίας των διαρθωτικών ταμείων και την χρήση τους και την χρησιμότητά τους για τις ε, πληθυσμούς των τσιγκάνων από δύο προοπτικές. Από τη μια πλευρά είμαστε μια οργάνωση μη κυβερνητική της Ισπανίας και εργαζόμαστε για την κοινωνική ένταξη του πληθυσμού των τζιγκάνων και από το 2000 είμαστε ένας ενδιάμεσος διαμεσολαβητικός οργανισμός που αγωνίζεται κατά των διακρίσεων. Διαχειριζόμαστε άμεσα κονδύλια και με αυτήν βάση αυτή την εμπειρία έχουμε μπει και στο Euroma Network που είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ε, χώρες, συμμετέχουν χώρες που έχουν τις μεγαλύτερους ε, τσιγκάνικους πληθυσμούς, Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Σουηδία και η Πολωνία. Εργαζόμαστε από το 2007 έτσι ώστε όσοι διαχειρίζονται τα διευθυντικά ταμεία, η μονάδα δηλαδή διαχείριση των ε, κοινωνικού ταμείου, του Ευρωπαϊκού δηλαδή κοινωνικού ταμείου, για κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους. Και μέσα σε αυτό το δίκτυο εργαζόμαστε από το 2007 και θα ήθελα λοιπόν την παρουσίασή μου να σα ε, την παρουσιάσω μέσα στο... Μέσω μάλλον των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει και μέσω της ανάλυσης και των προτάσεων που έχουμε προετοιμάσει για αυτή την περίοδο προγραμματισμού και να ολοκληρώσω με μια πρακτική παρουσίαση για το τι είναι το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα και ένα παραπάνω παράδειγμα για τα προγράμματα τα οποία οδηγούν σε αλλαγές στον, στην περίπτωση του Ταμείου Συνοχής, της πολιτικής συνοχής μάλλον. Έχουμε λοιπόν ε, ένα δίκτυο για δύο κρατημέλη ε, τα τελευταία δύο χρόνια αναλύσαμε ποιες ήταν, ε, ε, ποια ήταν τα διδάγματα αυτής της περίοδου προγραμματισμού και η χρήση των διευθυντικών ταμείων για την ένταξη των τσιγκάνικων πληθυσμών και έτσι ώστε να προγραμματίσουμε καλύτερα την επόμενη προγραμματική περίοδο και θέλω να σας δώσω ποια είναι τα πιο βασικά και ξεκάθαρα μηνύματα παρότι έχουμε πολλές εκθέσεις και μελέτες. Πρώτο λοιπόν είναι ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Εδώ θα πρέπει να μπορέσουμε μέσω της ε, ε, ε, προτεραιότητας, επενδυτικής προτεραιότητας 9.2 να στοχεύσουμε στη συνένταξη των πληθυσμών Ρωμά. Με βάση το 9.2 προσπαθούμε να αποζημιώσουμε τις, ε, μάλλον αντισταθμίσουμε τα πλεονεκτήματα των ε, πληθυσμών αυτών, αλλά μην ξεχνάμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ε, καταπολέμηση της στόχης, πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρώπης 2020, ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και το στόχο 8, το θεματικό στόχο 8 και το θεματικό στόχο 10. Επίσης θα πρέπει κάθε φορά στους στόχους ε, να προχωράμε ε, και είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τους πληθυσμούς Ρωμά στα επιχειρησιακά προγράμματα. Εν γέννη μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα ωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Ως προς αυτό θα θέλαμε ο στόχος αυτός, το target αυτό να είναι απαραίτητο ε, για να πραγματικά να μπορέσουν να ωφεληθούν ε, και να ενσωματωθούν ε, όχι μόνο λόγω της εθνοτικής τους κατάστασης αλλά και λόγω των διακρίσεων από τις οποίες υποφέρουν μέσα στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής περίοδου. Να ενσωματωθεί δηλαδή ο πληθυσμός των Ρωμά και στα υπόλοιπα προγράμματα, τα, όχι μόνο αυτά που καταπολεμούν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Απ' την άλλη πλευρά θέλουμε να υπάρξει γενικευμένη χρήση των προγραμμάτων, ιδιαίτερα του Κοινωνικού Ταμείου, μέσω της καταπολέμησης της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 20% μάλιστα του προϋπολογισμού προορίζεται για αυτά τα προγράμματα. Όμως, ε, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης της Υπέθρου επίσης θα πρέπει να εντάξουν στους δικαιούχους τους πληθυσμούς Ρώμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από την πολιτική συνοχή και από τα διάφορα ταμεία και κονδύλια ώστε να μπορέσει να ενταχθεί ο πληθυσμός στο Ρωμά και όχι μόνο να ωφεληθούμε από το κοινωνικό ταμείο. Τομεί τώρα παρεμβάσεων. Έχουμε στοχεύσει περισσότερο στην ε, παιδεία, στην απασχόληση, είναι πιο πρόσφατο, αλλά και στην ε, κοινωνική και ε, κοινοτική ένταξη. Θέλουμε δε, να υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, στέγαση, όπως σας είπα προηγουμένως το FEDER, το οποίο συνδέεται και με την ε, κοινωνική συνοχή. Θέλουμε ε, και πιστεύουμε ότι έχει μεγάλο δυναμικό, παιδική φτώχεια, να δουλέψουμε με το φαινόμενο της μετακίνησης των πληθυσμών το Ρωμά, να έχουμε δηλαδή οριζόντιες δυνατότητες παρέμβασης. Ένα επίσης σημαντικό θέμα είναι ότι ότι οι οριζόντιες αρχές των ίσων ευκαιριών και των μη διακρίσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα. Έχει γίνει αυτό, αλλά δεν αρκετή στην πράξη δεν βλέπουμε από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αρχών της ισότητας ευκαιριών και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Όσον αφορά τον αντίκτυπο, αυτό που είδαμε σε αυτή την περασμένη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η πολιτική συνοχή και τα ιδιωτικά ταμεία χρησιμοποιήθηκαν ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες, δηλαδή βασικές υπηρεσίες για τους πληθυσμούς στο Ρωμά. Αυτό που λέμε κάποια ε, μέτρα τα οποία είναι ας πούμε ρυθμιστικά μια παρηγοριά ας πούμε. Δεν είναι πραγματικά όμως ε, μέτρα. Θα πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση, ορθή χρήση της πολιτικής συνοχής ως ένα μέσο ε, δυνητικό το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική ώστε να προωθηθούν διαρθρωτικές αλλαγές, δηλαδή κοινωνική προώθηση του πληθυσμού των Ρωμά. Δεν είναι μόνο η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών, αλλά και η κοινωνική τους ένταξη. Επίσης όσον αφορά τον αντίκτυπο, αυτό που προωθούμε είναι αυτό που είδαμε στη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου που υπήρξαν πολλές ε, παρεμβάσεις, όμως βραχυπρόθεσμες ή σε μικρή κλίμακα. Υπήρξε ένας κατακαιρματισμός πόρων και άρα ο αντίκτυπος των μέτρων των διευθυντικών ταμείων ήταν περιορισμένο. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι να ε, φροντίσουμε να γίνουν προγράμματα μεγαλύτερης κλίμακας, μεγαλύτερων διαστάσεων, ώστε να έχουν πραγματικά αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης και στην κοινωνική ένταξη των ε, πληθυσμών Ρωμά. Τώρα, ολοκληρωμένη η στόχευση και η κοινωνική ένταξη των Ρωμά σημαίνει πολυδιάστατη προοπτική. Θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένοι στόχοι όσον αφορά τις παρεμβάσεις, δηλαδή παιδεία, απασχόληση, στέγαση, υγεία, ε, αλλά σε αυτό σε συνδυασμό των ταμείων, κοινωνικό ταμείο, ΦΕΝΤΕΡ και Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου οι δυνατότητες που προσφέρουν ε, τα ταμεία για να μπορέσει κανείς να επενδύσει σε αναλύσεις και έρευνες είναι πολύ σημαντικοί για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε τους πόρους και τα μέτρα στις πραγματικές ανάγκες ε, των ε, Ρωμά. Επίσης πρέπει να έχουμε πληροφορίες για το πώς ε, έχει η κατάσταση των Ρωμά, πού βρίσκονται αυτοί, γιατί έτσι θα μπορέσουμε καλύτερα να προσανατολίσουμε τους πόρους, αλλά και να τους νομιμοποιήσουμε, διότι πολλές φορές ε, ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι για τους πληθυσμούς Ρωμά όταν γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει η κατάστασή τους, δικαιολογούμε και αιτιολογούνται μάλλον οι δράσεις μας. Ενώ πολλές φορές χρηματοδοτούνται από, το ίδιο, από τα ίδια τα διευθυντικά ταμεία έρευνες, χάρτες, ε, μελέτες για τις συνθήκες διαβίωσης των ε, πληθυσμών Ρωμά. Τώρα, η ανάλυση μας είναι ότι ο προγραμματισμός για την ε, ε, περίοδο εφαρμογής θα πρέπει να γίνει, να προχωρήσει περισσότερο. Η Ρωμά είναι πιο παρόντες στα επιχειρησιακά προγράμματα και όσον αφορά τον προγραμματισμό υπήρξε πρόοδος. Όμως αυτή τη στιγμή η μεγάλη πρόκληση είναι η εφαρμογή. Και ως προς αυτό το Κοινοβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ρόλο να παίξουν στην παρακολούθηση, στο να μας εξασφαλίσουν ότι αυτά που προγραμματίσαμε θα υλοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο και μέσα σε έναν ορίζοντα 2020-2023 η κατάσταση διαβίωσης, οι συνθήκες διαβίωσης θα έχουν βελτιωθεί ως αποτέλεσμα των επενδύσεων μέσω της πολιτικής συνοχής. Και τώρα θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα και είναι το πρόγραμμα το οποίο εμείς διαχειριζόμαστε στην πράξη από το 2012 ε, με, σε συνεργασία, από το 2000 ε, σε συνεργασία με το Διαθετικά Ταμεία. Να δώσουμε δηλαδή ποιε είναι οι προοπτικέ και ποιε είναι οι προσδοκίε. Οι προσδοκίε γενικά είναι χαμηλέ, ενώ υπάρχουν προγράμματα τα οποία λειτουργούν και προωθούν κοινωνικέ αλλαγέ. Στη δική μα ε, περίπτωση, το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταπολεμά τι διακρίσει στην Ισπανία ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πραγματικά πρωτοπόρο το 2000. Ε, σχεδιάστηκε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα όπου περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την κοινότητα των Ρωμά, αλλά όχι αποκλειστικά για αυτήν. Διάφορες ευάλωτες ομάδες βλέπετε εδώ, ισότητα των γυναικών, των, φίλων, άτομα με ειδικέ ανάγκες, μετανάστες κτλ. Και εκεί οι μηνότητε μέσα σε παρενθέσεις φαίνονται οι Ρωμά. Δηλαδή, ναι, είναι και αυτή η στόχη, αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ευρύτερο πρόγραμμα έχουμε και κοινωνικές μάλλον ε, μονάδες έτσι ώστε ε, να έχουμε ειδικευμένε μονάδες που έχουν μια συγκεκριμένη πορεία εργασίας και μπορούν να έρθουν πιο κοντά στις ε, στοχευμένες ομάδες. Και ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε σε δύο πλαίσια αυτό της απασχόλησης και αυτό της παιδείας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά παίζουν βασικό ρόλο για τις αλλαγές. Το πρόγραμμά μας ονομάζεται «Πρόσβαση» ε, και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορέσει να έχει πρόσβαση ο πληθυσμός Ρωμά στην αγορά εργασίας. Προωθούμε την κατάρτιση, διότι συνήθως δεν έχουν πολλές δεξιότητες, δεν έχουν πολλή εμπειρία και δεν έχουν επίσης ε, ε, συστάσεις γιατί συνήθως εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν είναι αναγνωρισμένες. Εργαζόμαστε με συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα πορεία, γιατί στόχος είναι η ισότητα των ευκαιριών, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά το σημείο εκκίνησης δεν είναι το ίδιο για όλους και άρα πρέπει με διαφορετικό τρόπο να επενδύσουμε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Δουλεύουμε με συγκεκριμένους στόχους, αλλά όχι αποκλειστικούς. Το 70% των δικαιούχων είναι Ρωμά. Είναι ένα ειδικευμένο πρόγραμμα για ε, Ρωμά, αλλά δεν είναι αποκλειστικά για Ρωμά. Το 30% είναι άνθρωποι που δεν είναι Ρωμά. Είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει τα αποτελέσματα και σε αυτό, μέσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μετράμε τα συμβάσει εργασία, δηλαδή όχι τι προηγούμενε φάσει κατάρτιση κτλ, αλλά τον αριθμό συμβάσεων που επιτυχάνουμε. Ανάλογα με το είδο επαγγέλματο, με συγκεκριμένη μεθοδολογία, ξεκίνησε ω πιλωτικό πρόγραμμα και τώρα έχει διευρυθεί σε εθνικό επίπεδο και συνεργαζόμαστε και μάλλον εφαρμόζεται σε 50 Δήμου τη Ισπανία. Είναι φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε κοινωνικέ αλλαγέ και αυτά εδώ είναι τα αποτελέσματα. Από το με μέχρι το 2014 είχαμε πάνω από 80.000 δικαιούχους και ο αριθμός των συμβάσεων που επιτύχαμε ήταν 58.000. Ο αριθμός των ανθρώπων που μπόρεσαν να έχουν σύμβαση Εργασία ήταν 22.561, ενώ το 53% εξ αυτών ήταν γυναίκες, γιατί έχουμε και δράσεις με προοπτική φύλου. Ε, συμμετείχαν πάνω από 3.000 εταιρείε σε αυτό το πρόγραμμα. Το αριθμός των καταρτήσεων ήταν 2.800 και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το 2014 που ήταν το τελευταίο έτος σε η κρίση οικονομική στο απόγειό τη και αυτά εδώ είναι τα στοιχεία μας. Ε, το 2014 καταφέραμε να έχουμε 5.000 συμβάσει εργασίας, συμβάσει απασχόλησης. Όσον αφορά τι κοινωνικέ αλλαγέ, έχει τεράστιο αντίκτυπο λοιπόν γιατί έτσι ο πληθυσμό των Ρωμά έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η πρόεδρο διακόπτη, συγγνώμη, σα ζητώ να ολοκληρώσετε. Δεύτερος άξονας είναι η ε, παιδεία και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου. Εργαζόμαστε με τους ε, σπουδαστές, με τις, με τις οικογένειες και τα κέντρα και θέλω να σας δείξω μόνο τα αποτελέσματα. Εργαζόμαστε με 1.357 μαθητές και καταφέραμε 524 να τελειώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αυτό είναι το τελευταίο μας μήνυμα, γιατί πραγματικά θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία λειτουργούν και πραγματικά όταν υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι κολλά προσανατολισμένα και ε, έχουν σωστά στοχεύσει τους ε, Ρωμά, έχουν αποτελέσματα και είναι επίσης σημαντικό να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό των ιδιωτικών ταμείων με στρατηγικό τρόπο ώστε να προωθήσουμε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις κοινωνικές και όχι μόνο για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες των Ρωμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που είμαι υποχρεωμένη να σας διακόψω, αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος. Uh, Έχω τη χαρά να δώσω το λόγο τώρα στην ε, δόκτωρα Φραντσίσκα Γκίφαη. Uh, ε, ζητώ συγγνώμη. Είναι δήμαρχος ε, του Νόικολν στο Βερολίνο. Έχετε το λόγο να μας κάνετε την παρουσίασή σας σε 10 λεπτά. So, ladies and gentlemen, good morning. Greetings. Καλημέρα σας. Χαιρετισμούς φιλιά από το Βερολίνο. Εγώ είμαι δήμαρχος ενός διαμερίσματος, ο δήμος λέγεται Νόικέρν. Ε, ορίστε, χαιρετίσματα από το Δημαρχείο που βλέπετε εδώ, εκεί εργάζομαι. Ε, ήθελα να σας δείξω λίγο το Βερολίνο. Είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, η πρωτεύουσα της Γερμανίας 12 είναι τα διαμερίσματα επιμέρους δημη Εδώ στο κόκκινο βλέπετε τον Όικολ που είναι ο δήμος μου. Έχουμε περίπου 300 μισό λεπτό να το βρω. Έχουμε 300.000 κατοίκους και πολύ πολιτισμική είναι η πόλη μας. Ε, περίπου ο μισός πληθυσμός ε, προέρχεται από τη μετανάστευση ε, είναι 60 ε, εθνότητες και τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε δεχθεί ιδιαίτερα κόσμο από το, τα Βαλκάνια, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, έρχονται στη Γερμανία, στο Βερολίνο και ιδιαίτερα στο δικό μας Δήμο και μάλιστα πολλές από τις οικογένειες αυτές είναι Ρωμά. Δεν είναι δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και έχουν υποστεί διακρίσεις. Έχουν έρθει εδώ λοιπόν για μια καλύτερη ζωή, θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και για τα παιδιά τους και για μας. Καμιά φορά αυτό η κατάσταση είναι πάρα πολύ ε, μεγάλη πρόκληση. Έχουμε περίπου 6.000 Βουλγάρους και Ρουμάνους ε, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι, καταχωρισμένοι επίσημα, αλλά υπολογίζουμε ότι ο πραγματικός αριθμός των μη εγγεγραμμένων είναι πολύ μεγαλύτερος. Πολλοί ζουν από κοινωνικά επιδόματα, ε, επίδομα τέκνων, επίδομα κοινωνικό, ε, προνοιακό, 40% ζουν λοιπόν από πόρους του κράτους και έρχονται να προσθεθούν σε μία πόλη που έχουμε ήδη πολλά προβλήματα. Έχουμε πάνω από 160 έθνη και 60 και 70% παιδική φτώχεια σε πολλές γειτονιές και δεν είναι εύκολο να έρχονται νέοι να προστίθενται που είναι οι ίδιοι σε πολύ επισφαλή κατάσταση και δύσκολη. Εκεί προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κονδύλια από εκεί. Έχουμε αντλήσει πόρους τα τελευταία χρόνια. Δύο διαφάνειες θα ήθελα να σας δείξω για να συνοψίσω λίγο τι έχουμε κάνει και τι στοχεύουμε. Oh, Great. So, I try again. προσπαθήσω και πάλι. We are using very... Ε, αντρούμε πάρα πολλά κονδύλια από το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, το ΦΕΝΤΕΡ, ε, για τη διαχείριση των διαφόρων γειτονιών. Έχουμε συνοικίες 11 ε, μεγάλες με κοινωνικά ε, προβλήματα και κοινωνική στέρηση και δίνουμε χρήματα για την ένταξη ε, και την κοινωνική συμπερίληψη. Την τελευταία προγραμματική περίοδο 2007-2013 αντλήσαμε περίπου 50 εκατομμύρια από ε, το ΦΕΝΤΕΡ και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε στους βασικούς τομείς που αναφέρετε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή στην εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, αγορά εργασίας. Αυτό το έχουμε όλοι από κοινού πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους τομείς και υποστηρίζω πάρα πολύ ε, τα όσα είπε η κυρία Φερνάντες, η προλαλήσασα. Δεν έχει νόημα δηλαδή να στοχεύουμε σε μία δράση ε, συγκεκριμένα για τους Ρωμά. Ε, πρέπει να γίνει μια συνολική δράση για όλο τον πληθυσμό που κατοικεί εκεί. Δεν είναι καλό για την κοινωνική ειρήνη, δεν προάγει την κοινωνική ειρήνη όταν στοχεύει σε δράσεις μόνο για τους Ρωμά σε μια δύσκολη περιοχή. I just tell you something. Θα ήθελα να σας πω τώρα μερικά πράγματα που κάνουμε στην παιδεία. Πολύ συχνά ε, διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά που έρχονται από οικογένειες Ρωμά, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία δεν έχουν ξαναπάει σχολείο. And very often... Ούτε γερμανικά μιλάνε και πολύ συχνά οι γονείς τους είναι αναλφάβητοι. Προσπαθούμε λοιπόν να οργανώσουμε στα σχολεία τάξεις υποδοχής. Έρχονται σε ε, ε, μικρές ομάδες για να μάθουν καν τη γλώσσα και να, προσπαθούν, να προετοιμαστούν για να παρακολουθούν κανονικά το σχολείο. Αυτό ε, στη δική μας πόλη, στο Δήμο μας έχουμε πάνω από 30 τέτοιου τάξεις και από τη ε, Βουλγαρία και τη Ρουμανία πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κάθε μήνα φτάνει μια σχολική τάξη σε αριθμό παιδιών. Ε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πάνω από 400 τάξεις υποδοχής υπάρχουν συνολικά ε, στην πόλη του Βερολίνου, στους 12 δήμους. Για τα ζητήματα υγείας τώρα, ε, το σημαντικότερο θέμα και ελπίζουμε να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι οι περισσότεροι που έρχονται είναι ανασφάλιστοι είναι ασφαλισμένοι ε, στη χώρα τους αλλά δεν πληρώνουν τις, τις εισφορές τους ε, και δεν καλύπτονται στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή στη Γερμανία. Αυτό το θέμα λοιπόν της υγειονομικής ασφάλισης και του εμβολιασμού. Είναι τα πιο οξέα προβλήματα. Επίσης, οι έγκυες και πολλοί νέες γυναίκες δηλαδή που είναι έγκυες είναι ανασφάλιστες και πάνε στα νοσοκομεία μας για να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Φοβούνται και πολύ συχνά μετά το τοκετό σηκώνονται και φεύγουν από το νοσοκομείο. Φυσικά κανείς δεν πληρώνει ε, τα έξοδα του και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Το τρίτος τομέας, τα, τα δύο πρώτα είπαμε ήταν η παιδεία και η υγεία, τρίτος μεγάλος ε, τομέας με οξέα επίσης προβλήματα είναι η στέγη. Έχουμε πολλές οικογένειες Ρωμά που φτάνουν ε, στο Βερολίνο και έχουν πρόβλημα να βρουν ένα κανονικό διαμέρισμα. Και υπάρχει και μία μπίζνα που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτό. Υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι που θεωρούν ότι α, ορίστε έρχεται τώρα μια οικογένεια που έχει οτι οριστε ερχεται τωρα μια οικογενεια που εχει προβληματα δεν μπορεί να βρει κανονικά διαμέρισμα. Οπότε σου δίνω ένα στρώμα, 200 ευρώ το μήνα και όταν βρεις διαμέρισμα, 20 τετραγωνικά, πληρώνεις 200 ευρώ το κεφάλι, οπότε καταλαβαίνετε πόσο αποδοτικό και κερδοφόρο είναι αυτό. Παίρνεις ένα ερείπιο, βάζεις όσους μπορείς και χρεώνεις τα στρώματα 200 ευρώ και τους εκμεταλλεύεσαι. Σε όλες τις μεγάλες γερμανικές πόλεις βλέπετε τέτοια σπίτια, υπάρχουν αυτοί και όλες οι μεγάλες πόλεις εξηγούν ότι έχουν τα ίδια προβλήματα. Προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε κάτι από πλευρά του Δήμου, γιατί δεν είναι καλό για την κοινωνική ειρήνη. Όταν έχεις ένα σπίτι που μπορούν να ζουν 50 άνθρωποι ας πούμε κανονικά και στεγάζονται 200. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τι κάνουμε λοιπόν με τα διορθωτικά ταμεία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας είναι να διαρκούν τα προγράμματα, πώς να το πω, ε, ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα, να μην σταματάνε, για να υπάρχει ένα ε, ελάχιστο διάρκειας για να μπορεί να τρέξει το πρόγραμμα και να, λειτουργήσουν και να αποδώσουν τα μέτρα. Το είπαν και οι προλαλήσασες με ενσωμάτωση, ένταξη και ολοκληρωμένη, αυτά τα τέσσερα να συνδέονται. Ε, υγεία, παιδεία, εργασία και στέγαση. Αυτά τα τέσσερα είναι αλληλένδετα και χρηματοδοτούνται φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω κάτι για τη νέα προγραμματική περίοδο, ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα για την ένταξη στην αγορά εργασίας που είναι και στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου. Στη νέα προγραμματική περίοδο έχουμε το εξής πρόβλημα. Οι κανονισμοί και οι ρυθμίσεις είναι πιο αυστηροί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την μέτρηση της επιτυχίας. Και πολύ συχνά γίνεται μια συζήτηση και, και, ερώτηση Πότε επιτυχάνει ένα πρόγραμμα, ένα έργο, ένα σχέδιο. Όταν φέρνει τον κόσμο στην αγορά εργασίας. Αλλά με τις ομάδες που έχουμε εμείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις φέρουμε μέχρι την αγορά εργασίας. Εμείς αρχίζουμε από το μηδέν. Πρέπει να φροντίσουμε αυτές τις οικογένειες, τα παιδιά να πάνε σχολείο, οι άνθρωποι να φύγουν από αυτά τα ερήπια που ζουν. Δηλαδή δεν έχουμε την ίδια φετηρία όλοι η κανονική υποστήριξη μιας οικογένειας δεν ξεκινάει για μας από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ε, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Έχει μεγάλη σημασία ποιους δείκτες εξετάζεις. Και λες το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μάλιστα θα πρέπει να ε, επικεντρώνεται στην πραγματική εργασία. Με εδώ έχουμε άλλα προβλήματα και η Ρωμά συγκεκριμένα πολύ συχνά δεν μπαίνουν καν στην πρώτη αγορά εργασίας. Πρώτα πρέπει να τους εκπαιδεύσεις. Πολλοί, ας πούμε, ε, είναι αναλφάβητοι, δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση, όχι μόνο γερμανικά, ούτε την ίδια τους τη γλώσσα δεν μιλάνε της χώρας. Ξέρω εγώ, ισπανικά ή μια άλλη γλώσσα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε, να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και επίσης χρειαζόμαστε χρήματα και ε, προγράμματα για ε, πολιτιστικούς διαμεσολαβητές, κοινωνικούς λειτουργούς, προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και για το κόστος διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών. Θα πρέπει να το σκεφτεί και να εστιάσει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Και επίσης διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τάση. Ορισμένα ΜΚΟ ή ορισμένοι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά τα προγράμματα προσπαθούν να επιλέγουν λίγο τους στόχους και τις ομάδες στόχους γιατί επειδή μετράνε την επιτυχία τους με τον αριθμό των ανθρώπων που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, επιλέγουν ποιους θα εντάξουν στο πρόγραμμα για να εμφανίσουν ότι έχει επιτυχία το πρόγραμμά τους. Οπότε δεν ασχολούνται με αυτές τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Εκεί θα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι φέρνουν μαζί τους όταν έρχονται και πώς έχουμε να κάνουμε πριν τους εντάξουμε στην αγορά εργασίας. Και εγώ έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Uh, Σταματώ εδώ σε πρώτη φάση και ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ελίζα Ονίλ Ρόγαν, που είναι αναπληρώτρια διευθύντρια για την εκμάθηση και τη συμμετοχή στο θέατρο Octagon στο Μπόλτον του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχετε το λόγο. Το Μπόλτον είναι μια πόλη στην Βόρεια Αγγλία με 276.800 κατοίκους. Από τον πληθυσμό αυτό 11,3% δεν έχουν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 13% εθνικά, σε εθνικό επίπεδο, 6,2% είναι γεννημένοι στην Ασία, 2,8% στην Ινδία, 1,8% στο Πακιστάν, 2% στην Αφρική, 1,3% στην Ανατολική Αφρική, το Μπόλτον είναι από τις ε, τοπικές ε, αρχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προστασίας ε, και έχουμε περίπου 100 πρόσφυγες που έχουν επαναγκατασταθεί, που κάθε χρόνο επαναγκαθίστανται στο Μπόλτον. Το Μπόλτον είναι μια ε, πόλη με υψηλά επίπεδα ανεργίας και φτώχειας, ε, μορφή πολιτιστική ε, διάσταση και σε μερικές περιοχές ε, ο λευκός ο βρετανικός πληθυσμός ε, επίσης έχει νιώσει μια περιθωριοποίηση. Υπάρχουν θέματα κοινωνικής συνοχής λοιπόν, αλλά υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των κοινοτήτων και αυτό οδηγεί σε απομόνωση. Έχουμε υψηλό επίπεδα φτώχειας που πολλές φορές οδηγούν σε έλλειψη εμπιστοσύνης για τις νέες κοινότητες κοινωνικές κατοικίες, οι ε, κοινωνικές αιστείες ε, ε, μερικές φορές περιορίζονται σε συγκεκριμένες συνοικίες και τα διαχειρίζονται ιδιωτικά μεσητικά γραφεία. Βέβαια, έχουμε στερή συνεργασία με το Bolton at Home που είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που προσφέρει κοινωνικές κατοικίες. Το Μάρτιο του 2011 μετά από μια ψηφοφορία των ε, ε, ενοικιαστών ανέλαβαν ε, την κυριότητα των κατοικιών και αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται και έχουν την κυριότητα 18.000 κατοικιών. Προσπαθούμε να δώσουμε δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα που δημιουργούνται στις συνοικίες και στις κοινότητές μας. Μερικές φορές μιλούμε για πρόσβαση σε πολιτιστικές ευκαιρίες και αυξημένη συμμετοχή σε σχέδια, σε προγράμματα, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να μαθαίνει ε, για τη δική του κοινότητα, για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες κοινότητες και για τη θέση του στον κόσμο. Και χρησιμοποιούμε μια πολιτιστική προσφορά για να μπορέσει ο κόσμος ε, να αναπτύξει το πώς ε, νιώθει για πράγματα που θεωρεί σημαντικά, για θέματα κοινωνικής συνοχής, συνοχής των κοινοτήτων. Επίσης τα προγράμματά μας στηρίζουν τις κοινότητες προκειμένου να μεγαλώσουν μαθαίνοντας. Και μάλιστα έχουμε και πλατφόρμες που παρέχουμε στις κοινότητες για να ε, δημιουργήσουν οι ίδιες τις αλλαγές. Και μάλιστα δημιουργούμε και δυνατότητες διαλόγου, όχι μόνο μέσω των μελών, αλλά και μεταξύ των κοινοτήτων. Και πολύ συχνά το θέμα είναι η διαφάνεια. Ε, νιώθουμε ότι επενδύουμε στον κόσμο που αισθάνεται έτσι καλύτερα ε, στην καθημερινότητά του. Και οι δύο έχουν κοινή διαντολογία και στόχος μας είναι η χειραφέτηση των κοινοτήτων η συνεργασία των πολιτών ε, και η συζήτηση ε, θεμάτων κοινωνικής ε, αναζωογόνησης και αναζωογόνησης των κοινοτήτων. Οι περισσότεροι, ακριβώς επειδή ζουν σε αυτές τις κοινότητες, έχουν πολύ πιο ε, σημαντικές ε, σχέσεις και πολύ πιο αυθεντικές και εγνήσεις σχέσεις με τους κατοίκους αυτής της κοινότητας. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τέτοιες ικανότητες, ε, να καταργήσουμε φραγμούς, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην παιδεία, σε νέες κοινέ εμπειρίες, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για αυθεντικές σχέσεις από ανθρώπους με, με διαφορετική ιστορία. Επίσης έχουμε και βραχυπρόθεσμα προγράμματα, για παράδειγμα με μία ομάδα από γυναίκες της Σομαλίας και του Σουδάν. Στο σχέδιο αυτό έχω, φέραμε κοντά δύο κοινότητες για να συζητήσουμε το θέμα του ακροτηριασμού γενε, ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων στο Μπόλτον. Είναι ένα πολιτιστικό ζήτημα που ε, έχουν φέρει οι κοινότητες ε, στις παραδόσεις τους και μάλιστα γίνονται τέτοιες επεμβάσεις και στο Μπόλτον. Τώρα έχουμε φωνές που ορθώνονται και θέλουν να βοηθήσουν τις κοινότητες να σταματήσουν αυτή την πρακτική. Μάλιστα έχουμε δημιουργήσει και ένα θεατρικό έργο για να χειραφετήσουμε τις γυναίκες και να τις επιτρέψουμε να θέσουν αυτό το ζήτημα στις κοινότητές τους. Το θέμα δηλαδή του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα ακόμη και στον Πόλτον. Μάλιστα προβλήθηκε αυτή η ταινία, ε, αυτό το έργο μάλλον το θεατρικό και σε μια διεθνή διάσκεψη. Και θεωρούμε ότι τέτοιες λύσεις θα πρέπει να βρεθούν από την ίδια την κοινότητα, όχι ε, από επιταγές της αστυνομίας ή της ε, ε, Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας. Έτσι, θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να καταλήξουν σε μια κοινή προσέγγιση. Κάτι που σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να νιώθουν ντροπή για τα έθιμά τους. Πρόκειται για ένα θέμα που δημιουργεί απομόνωση και μυστικότητα μεταξύ των κοινοτήτων. Η δημιουργική όμως διαδικασία επιτρέπει στις ομάδες να καθίσουν και να συζητήσουν από εκείνο τα θέματα. Ήταν μια σύντομη παρέμβαση του θεάτρου αυτού, αλλά ακριβώ επειδή συνεργαζόμαστε και με την φιλανθρωπική οργάνωση, τον Bolton at Home, συνεχίζουμε έτσι το έργο στι κοινότητε αυτέ. Ένα παράδειγμα ενό πιο μακρόπνο σχεδίου είναι μια γυναική ομάδα που ε, ασχολείται με ένα δημιουργικό σχέδιο που αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, οι γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο προέρχονται από διαφορετικές κοινότητες. Ε, Έφτιαξαν ένα θεατρικό έργο και μια ταινία με θέμα ακριβώς την ενδοοικογενειακή βία. Και ακριβώς επειδή ε, συνεργάστηκαν χάρη στο σχέδιο αυτό, εδώ και ένα χρόνο έχουν δημιουργήσει και άλλες ομάδες άλλων κοινοτήτων. Έχουν δηλαδή ε, παρατείνει το σχέδιο και συμπεριλαμβάνουν κόσμο από διαφορετικές κοινότητες. Είναι μια πολύμορφη ομάδα και μάλιστα η ομάδα αυτή ζήτησε και εξωτερική χρηματοδότηση. Έτσι δημιουργούμε ένα μοντέλο βιώσιμο που δεν αποκλείει κανέναν και που θα γίνει υπότιμο και για άλλες κοινότητες. Μάλιστα, κάποιος που μετακόμισε από το Λονδίνο στο Μπόλτον και εργάζεται 12 χρόνια, πρόσφατα είπε ότι μόνο μετά τη συμμετοχή του σε αυτή την τελευταία ομάδα ένιωσε ότι το Μπόλτον είναι πια το σπίτι της και δεν θέλει να ξαναφύγει. Για μας η, συνοχή των κοινοτήτων δημιουργεί ένα ασφαλή χώρο που φέρνει τον κόσμο κοντά ώστε να βρει κοινά ενδιαφέροντα. Και τα σχέδια του Θεάτρου Octagon και του Bolton at Home δημιουργούν αυτό το περιβάλλον εμπιστοσύνης, στήριξης και μάθησης. Έτσι ο κόσμος ε, φοβάται λιγότερο τις διαφορές και τέτοιου του σχέδια ενισχύουν τη συνοχή γιατί ακριβώς εμπλέκουν το σύνολο της κοινότητας. Γιατί μπορεί να ξεκινούμε με μια ολιγομελή ομάδα, αλλά οι συνέπειες ε, του προγράμματος ε, και το πολλαπλαστικό αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Έτσι προσπαθούμε να προβάλλουμε τέτοιε πρωτοβουλίε και να ενθαρρύνουμε και άλλου από την ευρύτερη κοινότητα είτε να παρακολουθήσουν τέτοιε πρωτοβουλίε είτε να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξή του. Έτσι γίνονται και αυτή η κοινωνία αυτή τη εμπειρία. Προσπαθούμε με διαφανή, ανοιχτό και ασφαλή τρόπο να προβάλλουμε αυτά τα σχέδια που δημιουργούν ευκαιρίες για τις κοινότητε να βρουν τις δικέ τους λύσεις και να ξεπίσουν αυτόν τον ασφαλή χώρο για να αναζητήσουν διαφορετικές λύσεις στα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρου με διαφορετική ιστορία, γιατί η συμμετοχή στην τέχνη είναι πολύ δυναμικό εργαλείο για την αλλαγή της νοοτροπίας. Και το Bolton at Home, αυτή η φιλοθεραπική οργάνωση, είναι ένα μοναδικό μοντέλο και με την εταιρική σχέση που έχει με το θέατρο Octagon, είναι ουσιαστικά η μόνη οργάνωση παροχής κοινωνικής κατοικίας ε, με ε, δημιουργικές πρωτοβουλίες που αφορούν με την τέχνη και με έναν πλούσιο προϋπολογισμό που αφιερώνει σε τέτοιες δημιουργικές καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες συμμετοχής των κοινοτήτων. Χάρη σε αυτήν την εταιρική σχέση έχουμε μια πιο θεσμοθετημένη συμφωνία και η φιλανθρωπική οργάνωση Bolton at Home έγινε από τους βασικούς σπόνσορες του θεάτρου Octagon. Μάλιστα αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε 20.000 λίρες το χρόνο από το Bolton at Home και έτσι ε, δίνουμε ε, ε, ετησίως 1.800 δωρεάν εισιτήρια για τις παραστάσεις μας. Μάλιστα έχουμε και πρωτοβουλή συνοχής με τη φιλανθρωπική αυτή οργάνωση. Η δωρεάν πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο δίνει ευκαιρία σε πολλοί κόσμο από την ευρύτερη περιοχή του Μάζεστερ να παρακολουθήσουν και να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες μοναδικές καλλιτεχνικές εμπειρίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονές μας για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες ε, παραγωγικές ε, παρουσιάσεις τους που έβριθαν παραδειγμάτων και καλών παραδειγμάτων και φυσικά μας ενδιαφέρει και εκτιμούμε ιδιαίτερως ότι γίνεται αυτή η κοινή συζήτηση των προβλημάτων και θα δώσω το λόγο σε προενήγηλα στην συντάκτρια της έκθεσης, την κυρία Ρέντκε, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κυρία Ρέντκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομιλήτριες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις σας και πολυδιάστατες για το πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτό του είδους τα θέματα. Αυτό που κρατώ από σας, κυρία Κράστεβα, είναι η ανάγκη για καινοτομία στην κοινωνία Επίσης, στο σχέδιο έκθεσής μας το τονίσαμε αυτή την ε, ιδέα της συνεργασίας ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τις αρχές, ώστε να καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση κάποιων κοινοτήτων. Από εσά, κυρία Φερνάντε, ε, κρατώ περισσότερο το πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια προσέγγιση ενταγμένη σε όλε τι πολιτικέ, δηλαδή να έχουμε μικρέ στοχευμένε ε, μελέτε ή προγράμματα. Κυρία Κίφε, από εσά κρατώ το θέμα της μακροπρόθεσμης διάρκειας των προγραμμάτων. Είναι κάτι που τακτικά συζητάμε εδώ στην Περιφερειακή Επιτροπή και πώς θα δημιουργήσουμε στρατηγικές για ένταξη μακροπρόθεσμα. Και εσείς κυρία Χόγκαν τονίσατε σαφώς πιστεύω το πολύ σημαντικό μέσο του πολιτισμού και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα από τα εργαλεία για να περιλάβουμε, να εντάξουμε τις περιθωριοποιημένες ε, κοινότητες και θα πρέπει να το ξεχνάμε και όταν μιλάμε για πολιτική συνοχή. Πιστεύω ότι στην εργασία που κάναμε σε αυτό το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης γιατί είχαμε ήδη κάποιες συζητήσεις επί τη βάση των ε, ε, εγγράφων εργασίας. Πάντως συχνά όταν μιλάμε για περιθωριοποιημένες κοινότητες ε, φαίνεται λες και αυτές οι κοινότητες είναι το πρόβλημα. Ενώ ε, στις συζητήσεις που κάναμε εμείς καταστήσαμε σαφές ότι δεν είναι οι άνθρωποι που είναι το πρόβλημα, όχι οι περιθωριοποιημένες ε, κοινότητες, αλλά η δομική, διαρθωτική, ε, ο διαρθωτικός αυτός αποκλεισμός που αντιμετωπίζουν. Όπως στη Βουλγαρία, ας πούμε, βλέπουμε ότι η κοινότητα των Ρωμά δέχεται επιθέσεις ή άλλες ομάδες της κοινωνίας επιτίθεται και πολύ συχνά αυτά τα προβλήματα διαρθρωτικού αποκλεισμού βασίζονται σε διαφόρων ειδών ρατσισμούς και εμείς ως ομάδα θέλουμε να δούμε πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μέσα για την καταπολέμηση αυτού του διαρθρωτικού αποκλεισμού. Νομίζω ότι στη συζήτηση μέχρι στιγμής επίσης με την κοινωνία των πολιτών και εμπειρογνώμονες που έδωσαν πολλές χρήσιμες απόψεις διαπιστώσαμε, βρήκαμε μάλλον διάφορα σημεία εισόδου που η πολιτική συνοχή μπορεί να είναι ε, ακριβώς ένα εργαλείο για να καταπολεμηθεί η ο διαθωτικός αποκλεισμό και το πρόβλημα τη της διάκρισης εναντί περιθωριοποιημένων ε, κοινοτήτων. Αυτό ήδη έχει ενσωματωθεί στον κανονισμό του 2010 και στη νέα χρηματοδοτική περίοδο αποτελεί και πάλι μία από τις προτεραιότητες σε συμφωνία με τις ε, διεκδικήσεις των Ρωμά. Θα πρέπει να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί και τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον να δούμε ποιες προτάσεις μπορούμε να υποβάλουμε ώστε να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο όλα αυτά. Κάτι που συζητήσαμε επίσης ε, μακρόν με τους κοιόδες εισηγητές ήταν το θέμα του ορισμού. Δίνουμε ένα κατάλογο περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, δίνουμε ε, τα ανθρώπους με τις ε, αναπηρίες ε, ή κάποιοι, ομαδοποι, κάποιες ομάδες. Γιατί, τελικά είπαμε πως όχι γιατί ο κατάλογος ήταν πολύ μακρύς ε, ε, και δεν θα ήταν και πολύ χρήσιμος για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πολιτικές συνοχής για να καταπολεμηθεί ο διευθυντικός αποκλεισμός. Ε, είδαμε λοιπόν από την αρχή τον διορθωτικό αποκλεισμό, να δούμε ποιες ομάδες υποφέρουν από αυτό και πώς μπορούμε μέσω των πολιτικών που έχουμε να το καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Θέλουμε και η κυρία Φερνάντες, και, ε, η κυρία Φερνάντες μάλλον το τόνισε αυτό στην εισηγησή της, να δούμε πώς μπορούμε από την φάση του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και μέχρι την παρακολούθηση και την αποαξιολόγηση, να δούμε πώς μπορούν καλύτερα να ενταχθούν οι διάφορες ομάδες αυτές στις πολιτικές συνοχής και να καταπολεμηθεί κατά αυτόν τον τρόπο ο διαρθωτικός αποκλεισμός. Όταν βλέπουμε την πρώτη φάση, την προπαρασκευή και τον σχεδιασμό, προγραμματισμό ε, μέχρι στιγμής στις διάφορες ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης και στα επιχειρησιακά μας προγράμματα αναφέρονται ρητά αυτές οι περιθωριοποιημένες κοινότητες ε, αλλά Ήδη δηλαδή αντιμετωπίζονται στα προγράμματα τα βασικά για το θέμα του, ε, της περιθωριοποίησης, αλλά εμείς θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη στόχευση και ζητήσαμε την, ε, από την Κομισιόνα να, το, να μεριμνήσει εντονότερα γι' αυτό. Δεύτερη φάση στην προπαρασκευαστική, όταν εξετάζουμε την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, θέλουμε να δούμε ποιε αρμοδιότητε θα έχουν οι τοπικέ αρχέ. Ακούσαμε και από το τοπικό επίπεδο πολλά ότι δηλαδή λόγω έλλειψης γνώσης αλλά και επίσης λόγω έλλειψης ε, ευαισθησίας προέκυπταν προβλήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι στόχος μας να, ε, να θέσουμε και να δώσουμε βοήθεια στον κόσμο στις τοπικές αρχές ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ώστε να έχουμε ε, καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τώρα, εφαρμογή των προγραμμάτων, κάτι που ήδη ανεφέρθη επανελειμμένα, είναι το θέμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Να δούμε δηλαδή πώς στους διάφορους τομείς όπου οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες και όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ταμεία, να έχουμε δηλαδή πολυταμιακή <laughs> προσέγγιση, να, δηλαδή όχι μόνο το κοινωνικό ταμείο αλλά και άλλα ταμεία, όπως ας πούμε η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, πώς χρήματα δηλαδή από εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέους από τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, να δούμε την ατζέντα ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και η κυρία Κίφε μας έδωσε πολλές, μια πολύ καλή εικόνα. Στις αστικές περιοχές λοιπόν όπου υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις και πώς ε, ε, το θεματολόγιο για τις αστικές ε, περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η κατάσταση ολοκληρωμένη προσέγγιση μαζί με μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική που μάλλον θα είναι μεγάλη πρόκληση και επίσης στην εφαρμογή μια από τις προτάσεις που διατυπώνουμε στην έκθεσή μας είναι να ενισχύσουμε την, την οικοδόμηση δυνατοτήτων γιατί στο παρελθόν επανειλημμένα είδαμε ότι έλειπαν δυνατότητες και γι' αυτό και η αρχή της εταιρικής σχέσης δεν εφαρμόστηκε συχνά γιατί ο κώδικας συντολογίας δεν ήταν γνωστός ή δεν υπήρχε κοινωνία της ένταξης ε, και όσον αφορά την ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην ίδια την εφαρμογή των προγραμμάτων υπήρχε πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία τονίζουμε στην έκθεσή μας, ότι δηλαδή η ειδική της κατάστασης για το πώς θα καταπολεμηθεί η ο διαρθωτικός αποκλεισμός είναι ακριβώς ο κόσμος από αυτές τις κοινότητες. Και θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνονται, ε, να, εμπλέκονται μάλλον στην ε, σύσταση, σύνταξη των προγραμμάτων και στην επιλογή του πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα. Τελευταίο σημείο η αξιολόγηση έχει ήδη αναφερθεί πιστεύω όχι ίσως ρητά, αλλά το να έχουμε νούμερα, να έχουμε ποσοτική αξιολόγηση και κατά πόσο αυτό δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, το πρόβλημα του streaming ανεφέρθη ότι δηλαδή οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι κοινότητες, αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, ε, δεν είναι αυτοί οι οποίοι ε, επηρεάζονται από τα προγράμματα, αλλά αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας, δυναμικό επιτυχίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν να συνδυάσουμε τα στοιχεία, τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά. για να δούμε τις διάφορες διαστάσεις του προβλήματος στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Στη χθεσινή συζήτηση με, τον, με την Επίτροπο Τάισεν για το Κοινωνικό Ταμείο, η Επίτροπος είπε ότι για την ώρα η Κομισιόν εργάζεται πάνω στη σύσταση νέων δικτών. Είπαμε ότι θα πρέπει αυτοί να εστιάσουν, αλλά ίσως και εκπρόσωπος της Κομισιόν θα μπορούσε να μας πει δύο πράγματα. Και για να κλείσω, κάτι το οποίο σκεφτήκαμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την χειραφέτηση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων είναι να έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο. Ο κόσμος να μπορεί να συναντηθεί, να μπορούν να ανταλλάξουν καλύτερες πρακτικές και σήμερα ε, ακούσαμε για πολλές καλές πρακτικές γιατί έτσι μπορούν να μάθουν οι μένα από τους δε και να αλληλοβοηθηθούν για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Και γι' αυτό το λόγο, και ήδη αναφέρατε Πρόεδρε, θέλουμε να ξεκινήσουμε με αυτό το, τη δικτύωση να μην το αναφέρουμε μόνο στην έκθεσή μας, αλλά να το ξεκινήσουμε ήδη. Θέλω να σας καλέσω λοιπόν στη μεσημεριανό γεύμα δικτύωσης, όπου θα συμμετέχουν όλοι όσοι μας στήριξαν στη σύνταξη της έκθεσης μετά το τέλος της συνεδρίσης, γιατί πιστεύω μπορούμε να μάθουμε πολλά από αλλήλους και έτσι η πολιτική συνοχή να λειτουργήσει καλύτερα υπέρ των περιθωριοποιημένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρέντχε. Ε, αρχίζει τώρα η συζήτηση των μελών και αρχίζουμε με τους και ηγητές. Ο κύριος Γιάκοφ ήθελε το λόγο, ο κύριος Τσέλερ και μετά οι υπόλοιποι ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τις καλεσμένες που παρουσίασαν τις ιδέες, τις προτάσεις και τις εμπειρίες τους, τα βιώματά τους και που μας παρουσίασαν ε, κάποιες λύσεις που βρήκαν κοινότητες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά, αλλά και πώς μπορούμε να προτείνουμε τρόπους συνεργασίας διακοινωτικούς. Πολύ καλή πρωτοβουλία, αξιέπαινη και πολύ αξιόλογη. Είμαι υπέρ αυτής της προσέγγισης και είμαι υπέρ του τρόπου με τον οποίο χειριζόμαστε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας παραθέσω εδώ και, το και την προσωπική μου εμπειρία που μπορεί να ε, αποβεί χρήσιμη και για την ε, εισηγήτριά μας και θα μπορούσε ίσως να την ε, περιλάβει και στην έκθεσή της. Ε, τρεις είναι οι βασικοί άξονες. Σίγουρα είναι σημαντική η παιδεία, η εκπαίδευση. Ας μην ξεχνούμε όμως μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, βρυφονιπιακή σταθμή για τα παιδιά των Αθηγάνων, για τα παιδιά των Ρωμά. Με αυτό το θέμα ασχολήθηκα ιδιαίτερα εγώ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ώστε από τη βρεφική, από την υπιακή ηλικία ε, τα παιδιά των Ρωμά να μπαίνουν σε περιβάλλον κοινωνιοποίησης ε, και να δημιουργείται έτσι ένα ομαδικό έργο με επισκέψεις, ε, με ταυτόχρονα δουλειά και με τους γονείς. Είναι εξαιρετική σημασία αυτή η προσπάθεια από την υπιακή ηλικία των παιδιών του Ρωμά. Γιατί πολλά παιδιά το ρομπά πηγαίνουν μόνο δημοτικό και πολύ σπάνια α, γυμνάσιο και λύκειο. Αλλά στην Ίστρα η κοινότητά μας είχε πολύ καλά αποτελέσματα και μάλιστα με πολύ περηφάνεια ένα παιδί Ρωμά ήρθε και μου είπε ότι έλαβε και πτυχίο πανεπιστημίου. Είναι σημαντικό λοιπόν σίγουρα το εκπαιδευτικό σύστημα και είναι σημαντικό να προβάλλουμε τέτοια επιτυχημένα παραδείγματα και παιδιά Ρωμά που καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μελών της κοινότητας Ρωμά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχαμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Ίστρια που είχε μια ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία προσκαλούσε μέλη της κοινότητας Ρωμά που ε, παρουσίαζαν τα προσωπικά τους ε, βιώματα αλλά και διάφορες εμπειρίες στην κοινότητα ή τα διάφορα ζητήματα που τους αποσχολούσαν. Πολύ σημαντική λοιπόν και η πρόσβαση των Ρωμά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση, στα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να προβάλλονται και με τέτοιο τρόπο τα μέλη των Ρωμά. Γιατί ε, είναι σημαντικό με την πρόσβαση αυτή όχι μόνο να ακούν οι ίδιοι Ρωμά τους ε, συμπολίτε του ε, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, αλλά και οι υπόλοιπε κοινότητε να ακούν παρουσιάσει και εμπειρίες και βιώματα ή προβληματισμού στο Ρωμά. Παιδεία λοιπόν, και σταθμή, πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεύτερον και τρίτον, δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων, γιατί οι Ρωμά έχουν εμπειρία με ε, μικρέ μικρές δουλειές, περίπτερα, σε ε, οπότε και εμείς στην Πούλα, στην Ίστρια, καταφέραμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να μπορέσουν να αυτοαπασχολούνται οι Ρωμά σε τέτοιες μικρές δουλειές. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το σύστημα να το αναγνωρίσουμε. Γιατί δύσκολα ένας Ρωμά θα πάει να απασχοληθεί σε μια βιομηχανία, γιατί Γνωρίζοντα την οτροπία των Ρωμά, νομίζω ότι προτιμούν τέτοιε μικροδουλειέ περισσότερο, μικρέ επιχειρήσει και κυρίω την αυτοαπασχόληση. Και ένα άλλο θέμα που δεν έχει σχέση με του Ρωμά αφορά κάτι που είπε η συγγήτρια ότι δεν θα ήθελε να ορίσει τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Αλλά νομίζω ότι ήδη ξεκινήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Θα δημιουργήσουμε μια νέα έννοια και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Εγώ διαπίστωσα ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τους μετανάστες, αυτούς που έχουν σοβαρά προβλήματα στην κοινότητα, ε, είτε είναι άστεγοι είτε όχι. Εγώ ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τους αστέγους και τα προβλήματα των αστέγων, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να τους συμπεριλάβουμε και αυτούς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή σε κάποιο άλλο υπάρχον πρόβλημα. Καλό είναι λοιπόν και με αυτό το θέμα να ασχοληθούμε το επόμενο δίμηνο και να βρούμε μια λύση για το πώς θα ορίσουμε τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Και αυτό ε, θα χρειαστεί και για τις ε, επακόλουθες ε, επίσημες διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιάκοφτσης. Εγώ έκανα λάθος που δεν σας περιόρισα χρονικά, δεν είπα πόσο χρόνο δικαιούται ο καθένας με κούλπα, εγώ φταίω. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έκανα λάθος και δεν σας διέκοψε, ούτε σας είπα από την αρχή πόσο χρόνο δικαιούστε. Θα θέλω παρακαλούσα όμως τους υπόλοιπους ομιλητές να είναι πιο σύντομοι και να περιοριστούν στο λεπτό, 1,5 λεπτό το πολύ. Ο κύριος Τσέλερ. 1,5 λεπτό. Λιγότερο. Είναι πολύ λίγο. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που μου ήρθαν εδώ και μας κατέθεσαν την εμπειρία τους και μας βοηθούν με τις συμβουλές τους. Ευχαριστώ και την κυρία Ράιντ και την εισηγήτρια για το σχέδιο της έκθεσής της. Είχαμε συμφωνήσει και προηγουμένως το θέμα των περιθωριακών ε, ομάδων να το δούμε γενικά, αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στην ένταξη των ε, Ρωμά. Εκεί ε, εστιάζουμε ε, και το συνδέουμε με την πολιτική συνοχής. Για μένα ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι συζητάμε για τους Ρωμά και θέλουμε κάτι να κάνουμε για τους Ρωμά. Οι Ρωμά τι θέλουνε. Και μάλιστα τους θεωρούμε ομοιογενή ομάδα, που δεν ισχύει. Είναι 11 εκατομμύρια άνθρωποι που ανήκουν στον πληθυσμό των Ρωμά στην Ευρώπη και ζουν σε διαφορετικές ομάδες, σε διαφορετικές συνθήκες, ε, σε φυλές, σε μεγάλες οικογένειες που έχουν διαφορές μεταξύ τους. Και ο τρόπος ζωής τους τις τελευταίες δύο γενιές έχει αλλάξει. Μπορείτε, και το λέω αυτό εξαιτίας πείρας, το γνωρίζω προσωπικά. Και έχει υποστεί πολλαπλές μεταμορφώσεις. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 50 μέχρι και του 70 έβλεπα ακόμα πολλούς Ρωμά Τέλη του 70 και αρχές του 80 είδαμε την αναγκαστική αφομίωση σε πολλά κράτη ε, ανατολικά, από τη Σλοβακία μέχρι τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η αναγκαστική όμως ε, αφομίωση τι σήμαινε. Έγινε μια απόπειρα να ε, εγκαταστήσουν σε πόλεις ανθρώπους που είχαν νομαδικό τρόπο ζωής, αλλά χωρίς να τους εντάσσουν στην κοινωνία. Τους είχαν εξωθήσει στο περιθώριο. Γι' αυτό χαρακτηρίζονται και ως περιθωριακές ομάδες. Είναι άνθρωποι που ανήκουν μεν στην κοινωνία μας, αλλά τους είχαμε σπρώξει στο περιθώριο στα κράτη αυτά. Οπότε αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί να ε, παραμένει σήμερα. Ήδη υπόθηκε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για τους Ρωμά από τα διάφορα ευρωπαϊκά διασωτικά ταμεία με καθόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί η ενσωμάτωση και ένταξή τους και οι δυνατόν στις χώρες που είναι πατρίδες τους ή στις περιφέρειες που είναι πατρίδες τους. Αν όλα αυτά δεν συνοδεύονται με μια πολιτική βούληση για το πώς θα εφαρμοστούν, δεν βοηθούν καθόλου. Όσα λεφτά και να δίνουμε ή προθυμία να βοηθήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται η πολιτική βούληση και η προθυμία να υλοποιούνται αυτά. Και το δεύτερο, πώς τους προσεγγίζουμε τους ανθρώπους, γιατί και εντός της κοινότητας Ρωμά υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν ε, οι βασιλιάδες των Ρωμά που είναι εκατομμυριούχοι. Παρ' όλα αυτά κρατάνε τα μέλη της φυλής και της οικογένειά τους σε απόλυτη φτώχεια και εξάρτηση. Ε, Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και ιδιαίτερα σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τη θέση της γυναίκας που είναι ε, πραγματικά μη προνομιούχα και θα πρέπει να ε, ανυψωθεί το κοινωνικό τους καθεστώς και τα στάνταρτ. Και θα πρέπει να ρωτήσουμε και τους ίδιους τους Ρωμά, θέλουν να αφομοιώνονται ή θέλουν να συνεχίσουν να ζουν με την παραδοσιακή τους μορφή, ε, την παραδοσιακή ζωή που έχουν και θέλουν να έχουν μερική μόνο συμμετοχή στην κοινωνία μας, όχι πλήρη αφομοίωση. Και η μερική συμμετοχή είναι να τους δίνουμε τις ευκαιρίες που έχουν όλοι οι υπόλοιποι στην κοινωνία. Και το πρώτο που σκέφτομαι εδώ είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, το δεύτερο είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αν αυτά τα δύο πράγματα δεν συνδυαστούν, δηλαδή και ο διάλογος με την ίδια την κοινότητα το Ρωμά, δεν κάνουμε τίποτα και μάλιστα με ηθήνοντες ε, ή με ανθρώπους που να έχουν ε, κατασταλαγμένη άποψη, να μας πούν τι θέλουν και οι ίδιοι. Αλλιώς πώς θα ενταχθούν. Είναι αναφυσβήτητο ότι ανήκουν στην κοινωνία μας και θα πρέπει να έχουν και την αντίστοιχη συμμετοχή. Και από εκεί και πέρα ε, θα δούμε και τα κονδύλια. Δεν αρκεί λοιπόν να δίνουμε χρήματα και μόνο. Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση και όσοι φέρουν την ευθύνη θα πρέπει να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους για να ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταμάτος, κυρία Δησηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ευχαριστήσω τις ε, προσκεκλημένες μας αλλά και την εισηγήτρια που τις προσκάλεσε. Ήθελα να υπογραμμίσω και να ρωτήσω στήριξη από τις σχεώδεις σε σχέση με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Γιατί άκουσα για επιχειρησιακά προγράμματα στη διάρκεια των εισηγήσεων. Σαν άλυπε η στρατηγική φάση, το σημαντικό βασικό κομμάτι δηλαδή, ώστε να μπορέσουμε μετά καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία. Μιλήσαμε πολύ για κατάρτιση επίσης. Εγώ ξεκινώ και από αυτή την άποψη, αλλά από άλλο η οπτική γωνία. συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και σχολικά προγράμματα εκπαιδευτικά. Για παράδειγμα, σε κάθε ε, σχολείο της Ευρώπης θα ήθελα, ονειρεύομαι, να υπάρξουν προγράμματα τα οποία θα συμμετέχουν τα παιδιά ε, από όλες τις κοινωνίες ε, που είναι περιθωριοποιημένες. Δεν μιλάμε μόνο για τους Ρωμά, αλλά και τους άστεγους και τους ανάπηρους. για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε τα όσα ισχύουν. Δηλαδή ο άλλος δεν είναι διαφορετικός. Ε, μέσα στο πλαίσιο των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων να μιλήσουμε δηλαδή για παιδεία ε, ε, αφομοίωσης, ένταξης ήδη από τα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη σκιώδη εισηγήτρια είναι η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τι τέσσερι ομιλήτρε για τη συμβολή του σήμερα. Δυστυχώ δεν νομίζω πω θα μα επιτρέψει ο χρόνο να μπούμε σε πολλέ λεπτομέρειε. Πάντω, αν μπορούσατε να μα δώσετε τι εισηγήσει σα, θα ήταν πολύ ε, βοηθητικό για μα. Επίση, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη σημαντική δουλειά που έκανε για το θέμα και συμφωνώ ότι η ευθύνη για αντιμετώπιση αυτή τη ανάγκη, τη ανάγκη ανάγκες δηλαδή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων βασικά επιβαρύνει τα κρατή-μέλη, αλλά αναφίβολα, ακούγοντας και τις συμβολές της δικές σας, υπάρχει και σημαντικός ρόλος για τα, τα, τα Ταμείο Συνοχής σε ε, συμφωνία με τις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής αφομοίωσης. Πράγμα το οποίο βέβαια αμφισβητώ, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον αλληλεγγύη εδώ μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο θέμα μετά τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Ενδιαφερόμαστε περισσότερο λοιπόν για τις περιοθεροποιημένες ε, κοινωνίες ε, άσχετα από τον αντίκτυπο στους πιο ευάλωτους της κοινωνίας και γι' αυτό και χάρηκα για την ε, εφαρμογή και την παρακολούθηση για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση προς τις αρχές του προγράμματος και αυτό το λέμε όλη μου την προσοχή ε, που έδωσα σε όλα όσα μας είπατε, ότι δεν θέλετε δηλαδή τα χρήματα να πάνε μόνο στις τομείς τους τρεις της παρέμβασης. Το σχέδιο έκθεσης λέει ότι μπορεί εφαρμογή, πρέπει η εφαρμογή να, ε, να, να αντιστοιχεί στα κριτήρια της αφομοίωσης, αλλά όχι μόνο σε αυτά για το 20% που στοχεύεται στην ε, φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού ταμείου. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται να, είναι, ε, να ισχύει αυτό στη Βόρεια Ιρλανδία, στη δική μου περιφέρεια, όπου ο υπουργό Φάρη που είναι αρμόδιος για τα κοινωνικά θέματα χρησιμοποιεί το ταμείο αυτό για να βουλώσει μια τρύπα που προκλήθηκε από τους Βρετανούς Τόρι, τους Βρετανούς συντηρητικού και προσπαθεί να βοηθήσει οργανισμούς που συνεργάζονται πολύ στενά αυτή τη στιγμή με, κοινωνία, με τις κοινότητες στο Ρωμά, με, με τους ανέργους. Αυτοί είχαν πρόσβαση στο Ταμείο, αλλά περικόπηκε λόγω των δημοσιονομικών περικοπών και αυτό είναι αντίθετο με το πνεύμα του Κοινωνικού Ταμείου. Και έτσι επανέρχομαι και καλωσορίζω την αναφορά στην έκθεση για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Έχω κάποιες προτάσεις και πρέπει να πω ότι θα βασιστώ και στα σχόλια τα οποία ήδη έγιναν όσον αφορά τους σημαντικούς ορισμούς γιατί Εκτιμώ ότι μπορεί να είναι ένας ευρύς ορισμός ο ε, όρος περιθωριοποιημένες κοινότητες, πάντως υπάρχουν συγκεκριμένες που πρέπει να αναφέρονται, όπως ας πούμε οι κοινότητες των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες. Ξέρω πώς γίνεται αναφορά στην έκθεση στους Ρωμά και το καλωσορίζω, αλλά ως κάποιος που έχει γεννηθεί, μεγαλώσει και ζει σε μια μειονεκτική αστική περιοχή στη Βόρεια Ιρλανδία, καλωσορίζω και την αναφορά στην αστική νέα γενιά και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι άνθρωποι που ζουν σε μεθοριακές ή απομονωμένες περιοχές συχνά περιοθεροποιούνται λόγω της γεωγραφικής τους ε, ε, θέσης. Αν έρχεσαι λοιπόν από Ρώμα, αν είσαι Ρωμά και ζεις και σε περιθωριοποιημένη αστική περιοχή, χαιρετίσματα. Είναι ένα θέμα ε, το οποίο πρέπει και αυτό να το αναφέρουμε. Κλείνω λέγοντας πως είναι μια πολύ θετική πρώτη έκθεση ε, προσβλέπω στη συνεργασία με την εισηγήτρια και τις ε, υπόλοιπους σκιώδες εισηγητές ώστε να τροποποιήσουμε και να ενισχύσουμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σε εγώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τζούλι Γουόρ τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Μαρία και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν και μας παρουσίασαν ε, τις απόψεις και ευχαριστώ την Τέρι Ρέντκε και τους και όλους που ασχολούνται με το θέμα. Η συνοχή είναι πολύ σημαντική για μας ε, και ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μείνουμε συσπηρωμένοι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς με τα μέτρα της λιτότητας που έχουν αποτύχει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή η ανάγκη της ενότητας ε, και της διαφύλαξης της. Είχαμε πολλά αισιόδοξα παραδείγματα καλών πρακτικών και δουλειά στη βάση και χαιρόμαστε. Θα πρέπει να προβάλλουμε αυτά τα παραδείγματα και να αξιοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Εγώ σκέωτη συγγήτρια ε, προβληματίστηκα ε, και βασανίστηκα από το πώς θα ορίσουμε τις ε, περιθωριοποιημένες κοινότητες, ποιους θα περιλάβουμε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το δίλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και συμφωνώ με πολλά από όσα ακούσαμε από τους προλαλήσαντες. Δεν θα τα επαναλάβω, ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε κατά τη συζήτηση, την επόμενη συζήτηση της έκθεσης. Θα ήθελα όμως να αναφέρω κάτι που είπε η πρώτη μας καλεσμένη για το πώς μερικές φορές οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται τις ευάλωτες ομάδες γενικώ. Και το φαινόμενο του άλλου ε, ε, έχει επιταθεί. Έχουμε έξαρση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, ε, έξαρση του μίσους, της έλλειψης ανοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά φαινόμενα. Και μάλιστα μερικέ φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης νομιμοποιούν τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Και χαίρομαι που κάποιος συνάδελφος ανέφερε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σίγουρα η Ρωμά ήταν ιδιαίτερος εκτεθειμένη σε ένα ιδιαίτερο είδος ξενοφοβίας και ρατσισμού και βρέθηκα στο στόχαστρο αυτής της έντονης ξενοφοβίας. Το θέμα δεν είναι πώς αξιοποίησαν ή πώς αφελήθηκαν από προηγούμενες πολιτικές οι Ρωμά. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα ε, λειτουργήσουν ε, καλύτερα αυτές οι πολιτικές και για άλλες περιθωριακές κοινότητες στο μέλλον. Άκουσα με χαρά την αναφορά στη σημασία που έχει η παιδεία. Σίγουρα η παιδεία έχει θεμελιώδη σημασία, κεφαλαιώδη σημασία και όχι μόνο η επίσημη τυπική παιδεία αλλά και η διαβιοκατάρτιση, η άτυπη παιδεία, η ε, δουλειά και με τους γονείς και μάλιστα ε, σε περιθωριοποιημένες κοινότητες ε, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για να νιώσουν και αυτές οι κοινότητες ότι δεν είναι αποκλεισμένε. Και η εμπειρία από το Octagon Theater στο Μπόλτον ε, μας έδειξε πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να χαρακτηρίσει, να προσδιορίσει τα προβλήματα και να τα μοιραστεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Και με τέτοιες πρωτοβουλίες με πιο μακρόπρο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα θα έχουμε πολύ πιο θετικό πνεύμα κοινότητας. Επίσης θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους Ρωμά και πάλι και την επιχειρηματικότητα αναφέρθηκε από κάποιον ε, προλαλήσαντα και το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Γενικώ οι φτωχές και περιθωριοποιημένες κοινότητες αλλά και κυρίως οι φτωχές κοινότητες, οι άποροι δεν κατασπαταλούν πράγματα. Δεν έχουν πολλά και γι' αυτό δεν τα σπαταλούν άδικα. Το είδαμε όμως, αυτή την κατασπατάληση την είδαμε ιδιαίτερα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε όλο και περισσότερο για την κυκλική οικονομία και να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει. Μάλιστα, πολλοί σε περιθωριοποιημένε κοινότητε και ιδιαίτερα Ρωμά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από εμά ε, την κυκλική οικονομία. Και σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση της νεολαία, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θετική εμπειρία των κοινοτήτων. Γιατί μερικές φορές είναι θύματα, αλλά πολύ συχνά έχουν ε, πολλά πράγματα να μας διδάξουν και εμείς πολλά να διδαχθούμε από αυτές τις κοινότητες. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το γύρο των ε, σκιωδών ομιλητών και έχω άλλους 7 γεγραμμένους στον κατάλογό μου για συμμετοχή στη συζήτηση. Αν όμως θέλετε να προλάβει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει δύο λόγια και να δευτερολογήσει και η συγκήτρια, μπορώ μόνο ένα λεπτό να δώσω στον καθένα. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Βανίστερόι. Ready now. δεν είναι έτοιμος. Είστε έτοιμος για ένα λεπτό. Έχετε ένα λεπτό κύριε Βανίστερόι. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα. Δύο ερωτήσει βασικά. Πρώτον για την ίδια την έκθεση. Η Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδοτεί. Έχει σημασία. Ακούσαμε τόσα πολλά για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γνωμοδοτεί η Κοινωνική Επιτροπή γιατί συνδέεται με πολλές από τις δραστηριότητες μας αυτό το θέμα. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα ε, για την απορρόφηση των χρημάτων. Γιατί ε, ένα από τα πρώτα σχόλια που ακούσαμε ήταν ότι διευθύνται πολύ περισσότερα κονδύλια από απορροφούν τα κράτη. Το είπατε κι εσείς ότι συμφωνούμε συμβάσεις ε, εταιρικής σχέσης, το άρθρο 12 το λέτε στην έκθεση, αλλά χωρίς αυτή την αναφορά. Μήπως λίγο να τους κατονομάσουμε, να τους ξεμπροστιάσουμε αυτούς. Γιατί όταν λέτε ότι κάποιοι δεν απορροφούν, ωραία και από εκεί και πέρα τι. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία για την τελευταία προγραμματική περίοδο και την τρέχουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βον. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια προς την Ελίζα από τον Μπόλτον και ευχαριστώ και την ίδια και τις υπόλοιπες ε, κυρίες. Πριν ε, έρθω εδώ είχα αυτοδιοικητική εμπειρία και πολλά από όσα άκουσα από τη Λίζα ε, μου είναι οικία και μου θύμισαν προηγούμενη δράση που είχα και εγώ εκεί. Ε, ε, ότι θα πρέπει να έρχονται οι πρωτοβουλίες από τα κάτω και όχι να επιβάλλονται. Ε, καμιά φορά είναι δύσκολο να συμμετέχουν οι ίδιες οι κοινότητες γιατί διστάζουν να εμπλακούν. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Η δημιουργία δυνατοτήτων σίγουρα, αλλά καμιά φορά δεν αρκεί αυτό. και δεν αρκεί να συμμετέχει μια επιμέρους κοινότητα, χρειάζεται και ευρύτερη κοινωνία. Και πολλές φορές υπάρχουν αντιστάσεις και όταν διαχειριζόμαστε τα προγράμματα θα πρέπει στο κάθε πρόγραμμα να βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα και όταν έχουμε καλές πρακτικές να διαδίδονται, να τις μοιραζόμαστε. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα, καλό θα ήταν να συνεχιστεί η συζήτηση. Κύριος Μπόγκοβιτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω και εγώ φυσικά την έκθεση αυτή. Αυτό το θέμα συνδέεται στενά με την πολιτική ε, απασχόληση και την εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και για τη Σλοβενία φυσικά με ε, την υπόθεση των Ρωμά. Δεν είναι ανταγωνιστικοί οι άνθρωποι και δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο πάρα πολύ δύσκολα στην αγορά εργασίας. Και πολύ συχνά αρνούνται κιόλα τι προσφορέ που του γίνονται. Διότι τα χρήματα που τους προσφέρουν είναι λιγότερα από τα προνοιακά επιδόματα που παίρνουν. Ε, και έχει σημασία να ε, προσέξουμε να μην εστιαζόμαστε πάντα στα δικαιώματα, να κοιτάμε λίγο και τις υποχρεώσεις. Άλλο θέμα είναι οι διακρίσεις αυτό φαίνεται και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, υποδομή, για την υποστήριξη της υγείας, της παιδείας κτλ. Θα πρέπει η εκπαίδευση να αρχίσει από την πολύ μικρή ηλικία, αλλιώς κινδυνεύουμε να χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Χρειάζεται λοιπόν ε, ένα συνδυασμό κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και από κρατικούς και περιφερειακούς πόρους. Το είπε και η συνάδελφος από το Βερολίνο. Είναι σημαντικότατο το θέμα της συνέχειας της χρηματοδότησης. Είναι επταετή τα προγράμματα και δεν μπορούμε να έχουμε ένα χρόνο λεφτά και του χρόνου να μην έχουμε. Ε, καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσματα χρειάζονται μέχρι και μια δεκαετία για να έρθουν. Ο κύριος Έθριτς, ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ βλέπουμε ένα εξαιρετικό μικρό κόσμο των θεμάτων που μας απασχολούν. Ορισμένοι ε, ε, εποφελούνται ε, από τη γενεοδορία της Προέδρου ή την καλή της ψυχή και μακρηγορούν και κάποιοι άλλοι πιέζονται και ε, έχουν ε, τα αποθυμένα και στεναχωριούνται. αυτό γίνεται και στην κοινωνία. Όταν κάποιοι επωφελούνται ή κάποιοι άλλοι δυσανασχετούν. Στη Βρετανία έχουμε μια καλή ένταξη. Ας πούμε έχουμε τους ΣΥΧ, τους Αγγλοασιάτες, εξαιρετικούς επιχειρηματίες εντάσσονται, σκληρά δουλεύουν, πληρώνουν τους φόρους τους και έχετε και κάποιους άλλους που επωφελούνται από τα προνοιακά ε, επιδόματα. Και μην αρχίζουμε να μιλάμε για την ετερότητα και τα λοιπά, να θυματοποιούμε τον κόσμο. Δώστε τους ίσες ευκαιρίες να ανθίσουν όλοι να αναπτυχθούν και από εκεί και πέρα θα λυθούν τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να εξηγήσω ότι έδωσα περισσότερο χρόνο και οδησηγητές. Γι' αυτό έμεινε μόνο ένα λεπτό για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Χέντμαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο πρακτικές πτυχές ε, του θέματος. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμότατα την κυρία Ρέντκε, την εισηγητριά μας, γιατί είναι πολύ ισορροπημένη η προσέγγισή της και συμφωνώ με τις αδερές γραμμές ε, της έκθεσης που μας παρουσίασε. Προσοχή, η διασταυρωμένη αυτή χρηματοδότηση που αναφέρει η έκθεση, για παράδειγμα 90 παράγραφος 2 του κανονισμού, έχουν κύρια σημασία για τέτοιου είδου προγράμματα ή σχέδια όπως αυτά που μας παρουσίασαν οι καλεσμένες μας εμπειρογνώμονες. Προσοχή. Ε, στο άρθρο αυτό με τις 8 προτεραιότητες ε, του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έβαλε ένα ε, κατόφλι μόνο 10% του κοινωνικού ταμείου που μπορεί να συνδυαστεί με το αναπτυξιακό ταμείο. Αλλά σε καμία περίπτωση δίνονται κίνητρα στους δικαιούχους ε, των προγραμμάτων να καταθέσουν προτάσεις για τέτοιου είδους τόσο απαραίτητα προγράμματα. Επίσης θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για αλλαγή προσέγγισης. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό να μην ε, πιστοποιούνται οι δαπάνες ε, σε προγράμματα που δεν έχουν χαρακτηριστικά εταιρική σχέση. Εγώ θα ήθελα να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και ίσως ε, στα προγράμματα που υπάρχουν ε, στοιχεία εταιρική σχέση να δημιουργήσουμε, ε, να δώσουμε μπόνους και εκεί που δεν υπάρχουν τέτοια ε, κίνητρα να αφαιρεθούν μία. Να έχουμε ένα σύστημα περισσότερο θετικό με, προ, με προσθήκη κάποιων αμορίων και μπόνους, σε περίπτωση που έχουμε τέτοιες ε, στοιχείες εταιρικε εταιρικές ε, σχέσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησα κάπως, αλλά είχαμε μία έκτακτη συνεδρίαση για τις συμβαστικές, πρωτοβουλ... τροπολογίες, γι' αυτό και άργησα. Αν έχουμε μια χώρα που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας της ε, πολιτικής ε, κοινωνικής ένταξης είναι η Τσεχία, η τσεχική δημοκρατία. Η χώρα αυτή έχει πολλά προβλήματα, δεν είναι βέβαια η μόνη, αλλά έχει ιδιαίτερα προβλήματα και ε, τα 25 χρόνια που ακολούθησαν την πτώση του κομμουνισμού, 300 γκέτο δημιουργήθηκαν στη Τσεχία. Αυτά τα γκέτο είναι τελείως απομονωμένα αποκλεισμένα και είναι η απόρρια μιας λαθασμένης πολιτικής. Μάλιστα ε, τώρα που έχουμε πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Ήμουν ε, αντιδήμαρχος μιας ε, μικρής πόλης και προσπαθήσαμε, πασχίσαμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία των γκέτο και να δώσουμε έμφαση στην κοινωνική ένταξη. Μόνο με μία πρόθεση κοινωνική ένταξη ε, θα αποσοβήσουμε τη δημιουργία γκέτο και μόνο να δημιουργήσουμε πρόσφορες συνθήκε διαβίαση και για τα μέλη της κοινότητα Ρωμά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα της γετοποίηση και τη περιθωριοποίησης στην τσεχική δημοκρατία. Είχαμε ακόμη και υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ντροπή για την χώρα μου. Ευχαριστώ.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 που ανέφερε και που έθιξε αυτό το ευρωπαϊκό θέμα. Είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πιστεύω πως κάθε χώρα ε, πρέπει να λάβει τις αποφάσεις τις ε, συγκεκριμένες για κάθε χώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να ανταλλάζουμε και τις καλές εμπειρίες. Εγώ ως πρώην δήμαρχος είχα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Η συνάδελφος ε, δήμαρχος του ε, της περιοχής εκείνης του Βερολίνου ε, θα, τα γνωρίζει όλα αυτά. Ε, τα ανέφερε κιόλας. Πρέπει όντως να καταρτιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για αυτές τις κοινότητες. Είτε πρόκειται για εκπροσώπους ε, δαφικών συλλόγων ή εκπροσώπους υπουργείων ή άλλων φορέων που ενδιαφέρονται. Κάποιες φορές θέλουν να βοηθήσουν οι άνθρωποι αλλά υπάρχουν νομικά κείμενα που αυτό το εμποδίζουν. Πρέπει να οργανωθούν συγκεκριμένες μαθήματα, κατάρτιση, να δοθεί το δικαίωμα στις τοπικές αρχές να λάβουν συγκεκριμένε αποφάσεις, για παράδειγμα για τους ανθρώπους που δεν έχουν χαρτιά, να έχουν χάσει ή που, δεν, έχουν άλλα προβλήματα ή δεν έχουν έσοδα. Ε, θα έπρεπε οι τοπικές αρχές να μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε στους άλλους έτσι ώστε να βελτιωθεί η πολιτική συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχουμε δύο από τη Γενική Διεύθυνση Επασχόλησης και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εξαιρετική ευκαιρία που γίνεται αυτή η συζήτηση και αυτή η έκθεση γιατί στην Κομισιόν τώρα ολοκληρώνουμε μια σημαντική προσπάθεια μεγάλης κλίμακας όσον αφορά το σύνολο των ταμείων συνοχής για την περίοδο μέχρι το θα ξεκινήσω με τους Ρωμά. Ξέρω ότι η συζήτηση αφορά όλες τις, ε, τις ομάδες, ε, αλλά ξεκινώ με τους Ρωμά. Μπορώ να σας δώσω τρεις βασικές αρχές των όσων προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε σε διάρκεια της περίοδου 2014-2020. Καταρχήν να συνδέσουμε πολύ περισσότερο το πλαίσιο πολιτικής που αναπτύσσεται, όπως γνωρίζετε από το 2010, με τη χρηματοδότηση και εσωτερικά στις task force τις οποίες ηγείται η DG δικαιοσύνη και έχουμε επαφές με τα εθνικά σημεία επαφής κτλ. Έπειτα το θέμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης είναι κάτι το οποίο εμείς διακηρύσουμε ε, και στις δικές μας υπηρεσίες, στους αρμόδιους για τις διαπραγματεύσεις, αλλά και στα κράτη-μέλη. Τρίτον, στρατηγική σύνδεση όχι μόνο με τη στρατηγική των Ρωμά. Ξέρουμε στους κανονισμούς έχουμε το μηχανισμό της εξάντε ερεσιμότητας, έχουμε συγκεκριμένες σχέσεις με τους Ρωμά, αλλά όπως τονίζει και η συγκήτρια έχουμε πιο συγκεκριμένα θέματα. Έγιναν συγκεκριμένες αναφορές για τη μείωση της στόχιας, έχουμε στρατηγική για την παιδεία, στρατηγική για την υγεία, που συνδέονται όλες. Αυτά για τη γενική προσέγγιση. Έχουμε εκδώσει διάφορες οδηγίες, κατευθύντηρες γραμμές, αναφορά στο πρώτη δελτίο ε, που ξεκίνησε το 2014 και πολλά από τα όσα αναφέρατε, το θέμα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διάφορα ταμεία, της ε, διάστασης, της ε, ανάπτυξης της κάθε κοινότητας. Τα έχουμε τοποθετήσει ως δυνατότητες και διάφορες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικούς συνδυασμούς για να τα καταφέρουν. Έχουμε ήδη κάνει δηλαδή χρήση αυτής της ε, στρατηγικής. Δεν νέο στοιχείο που είναι σημαντικό τον έφερε η συγγήτρια, Το θέμα της του διαρθωτικού αποκλεισμού ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε μάλιστα σήμερα παρουσιάζουμε στην ομάδα εμπειρογνωμόντων αλλού στις Βρυξέλλες ένα σημείωμα για τη χρήση των ταμείων για την αντιμετώπιση της παιδείας και των ειδικών διακρίσεων απέναντι στις περιθωριοποιημένες ομάδες. Θα έπρεπε αυτό τώρα κανονικά να είναι υπό εξέλιξη θεωρητικά αυτή τη στιγμή μαζί με τα κράτη-μέλη. Κάποια σχόλια τώρα για την έκθεση. Καταρχήν για το σημείο 3 γίνεται να αφορά στο κατά πόσο δίνουμε πληροφορίες αρκετά ώστε κανείς να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Ε, αυτό το κάνουμε για τη νέα περίοδο και θα επανέλθω όσον αφορά τη φάση εφαρμογής. Τώρα, όσον αφορά τα, σε τα στοχοθετημένα και και, και τα γενικά ε, ε, μέτρα αν θέλουμε συγκεκριμένα μέσα, αν θέλουμε παιδεία. Εμείς δεν φτιάχνουμε δομές υγείας, ας πούμε, ειδικά για κάποιες ομάδες, αλλά ε, θέλουμε να καλύπτουν και τις ανάγκες εκείνων. Ε, να πούμε να βελτιώνουμε την ισότητα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Εκεί που έχουμε στοχευμένα μέτρα η έκθεση αναφέρεται στο γεγονός ότι τροποποιήθηκε το ΦΕΝΤΕΡ ε, το 2010 ώστε να έχουμε περιληφθεί και η στέγαση των περιθωριοποιημένων ομάδων και έχουμε δώσει και στοιχεία σχετικά. Τα αποτελέσματα δεν είναι απαραίτητο πολύ ενθαρρυντικά είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά τα πράγματα και στο σημείο 3 ζητάτε ανάλυση. Ε, έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά από τα όσα αναφέρετε σήμερα το πρωί. Αν αναφερθείτε στις κατευθυντήριες γραμμές έχουμε και ένα τμήμα για τα διδάγματα που αποκομίσαμε. Μεταξύ αυτών το έχουμε εντοπίσει αυτό το ζήτημα. Σημείο 12 που αφορά την συμμετοχή των περιθωριοποιημένων ε, κοινοτήτων στις συμφωνίες εταιρική σχέσης. Και εκεί μιλάμε για τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ακριβώς αυτό κάναμε. Όσον αφορά την DG Regio, έχουμε εστιάσει τις εκθέσεις μας στις πέντε αυτές χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης όπου έχουμε μεγάλους πληθυσμούς Ρωμά και έχουμε και συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα. Χρησιμοποίησαμε το 2014 ως βάση για τις χώρες αυτές. Αυτή ήταν η προσέγγιση που ακολουθήσαμε. Και όντως πολλές ε, καλύπτονται τα θέματα μάλλον από το κοινωνικό ταμείο όσον αφορά την απασχόληση, για την παιδεία, την προσχολική ε, και αυτό καλύπτεται, προσπαθήσαμε δηλαδή και αυτό να το καλύψουμε. Ε, ξεπερνάμε δηλαδή το θεματικό στόχο 9 για το κοινωνική ε, ένταξη. Έχουμε βάλει και την παιδεία εδώ. Συμφωνούμε για το θέμα της παρακολούθησης. Έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα και ε, σκοπεύουμε να έχουμε μια ενεργή προσέγγιση στην παρακολούθηση των όσων έχουν ε, τοποθετηθεί εντός των προγραμμάτων. Η ανάλυση δηλαδή είναι σαφής και το θέμα αυτό είναι θέμα συμμετοχής και της κοινωνίας των πολιτών και τα και τα και είναι θέμα το οποίο προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε πολύ προσεκτικά. Πανέρχομαι τώρα στο θέμα των ορισμών. Είμαστε στην ίδια γραμμή με την εισηγήτρια. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν αναφερθεί. Ας ακούσαμε το παράδειγμα των μεταναστών, των αστέγων. Αυτό που θα πράξουμε λοιπόν είναι να κάνουμε μια μελέτη ώστε να επανέλθουμε στα επιχειρησιακά προγράμματα, να δούμε πού υπάρχουν θέματα, πού γίνονται οι αναφορές στις περιθωριοποιημένες ε, κοινωνίες, να κάνουμε και τις πρώτες συζητήσεις με τις ε, ε, με, με τους αρχές διαχείρισης. Και τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι το σημείο 23, όπου λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εκδώσει ανακοινωθέν ε, για να πει ότι όντως προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και την κάλυψη των περιθωριοποιημένων ε, κοινοτήτων. Αυτό υιοθετήθηκε στις 17 Ιωθενίου ε, φέτος. Είναι αιτήσια αυτή η διαδικασία και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για το τι θα πρέπει να γίνει στο περίοδο 2014 με 2000 2020 και φυσικά μπορούμε να σας δώσουμε το σχετικό έγγραφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καρόν τώρα. Σωστά είπα το όνομά σας. Μπορείτε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος για ε, το σκέλος που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τώρα. Το είπε και η συγγήτρια ότι θα πρέπει οι ενεχόμενοι να συμμετέχουν περισσότερο και οι σκιώδεις συγγητές. Και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε προβλέψει στον κανονισμό να προωθήσουμε την ενδυνάμωση των ε, εμπλεκομένων, των ΜΚΟ και των κοινωνικών εταίρων κυρίως, εξασφαλίζοντας τη σωστή χρηματοδότηση από πλευράς κρατών μελών, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε δραστηριότητες δημιουργίας δυνατοτήτων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, καθώς επίσης και στις μεταβατικές περιφέρειες. Αυτό είναι πάρα πολύ προσφυλές λοιπόν, σε εμά και ε, έχει σχέση με το σημερινό θέμα που μας απασχολεί. Για τους δείκτες επίσης αναφέρθηκαν κάποια ε, σημεία και πολύ σωστά το έκανε η συγγήτρια, στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχουμε κοινούς δείκτες ε, αποτελέσματος αλλά και κοινούς ε, δείκτες ε, μακροχρόνιους για τις περιθεροποιημένες κοινότητες και μεταξύ αυτών τους Ρωμά. Αυτά καλύπτονται και από τους κοινούς δείκτες τα στοιχεία. Αλλά προφανώς κάποια κράτη-μέλη έχουν επιλέξει να επικεντρωθούν στους Ρωμά. Και θα περιμέναμε από τα κράτη-μέλη να έχουν ειδικού δείκτες από εκεί και πέρα, δηλαδή να επαγρυπνούν και εκείνα. Επίσης, ε, κάτι που τόνισε και ο συνάδελφος, υπάρχει σύνδεση και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ενθαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη που έχουν μεγάλους πληθυσμούς Ρωμά να εστιάσουν σε προτεραιότητες επενδυτικές για να ε, προωθήσουν ε, την κοινωνικο-οικονομική ε, ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες επιλεγμένες. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για μια πάρα πολύ σύντομη ε, τοποθέτηση για να συμπεράνει. Έχουμε φύγει εκτός χρόνου και έχει έρθει ήδη ο κύριος Κέσλερ και μας περιμένει. Οπότε παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Θα είμαι, σας το υπόσχομαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συνεισέφεραν στη συζήτηση αυτή. Ήταν πάρα πολύ γόνιμη και καρποφόρα. Ευχαριστώ και τους ομιλητές και πάλι, τις ομιλήτριες καλύτερα, που έθεσαν το πλαίσιο της συζήτησης. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που προέκυψαν. Ένα σύντομο σχόλιο για τα διάφορα σημεία που ακούσαμε και σας υπόσχομαι θα τελειώσω. Αυτό που είπε ο ο Γιάκοφσιτς για την προβολή, την ορατότητα και την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι γεγονός, δεν το λέει η έκθεση, είναι πολύ σημαντικό και θα βρω χώρο να το γράψω. Για σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Τσέλα, να μην μιλάμε για τους Ρωμά, να μιλάμε μαζί τους. Τώρα δεν είχαμε χρόνο να δώσουμε ε, το λόγο στον κύριο Φράνς που εκπροσωπεί το ε, Ίδρυμα Χίλτεβα Λαγκρέντς που είναι ο ίδιος Σίντι, δηλαδή ε, από τις κοινότητες στη Γερμανία θα συμμετέχει αργότερα στην εκδήλωση δικτύωσης που θα έχουμε. Και παρακαλώ μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή με εκπροσώπους στο Ρωμά και τον ΣΥΝΤΗ διαφόρων κοινοτήτων που συμμετείχαν και στην εκπόνηση της έκθεσης. Για την κυρία Νταμάτο, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και πολύ σημαντικό. Δεν χρειαζόμαστε μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα για ανθρώπους από την κοινότητα το Ρωμά, αλλά χρειαζόμαστε και ε, από τις κοινότητες ε, ε, των πλειοψηφικών ομάδων. Ας υπάρχει ένας αντιτσιγκανισμός που δεν τον έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ ε, στα προγράμματα σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην διδακτέα Ήλ. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Άντερσον. Το θέμα της λιτότητας και ιδιαίτερα εκεί που χτύπησε η κρίση Ε, και σας ευχαριστώ για τα ειδικότερα παραδείγματα και για την κυρία Ward που μιλήσε για τις βέλτιστες πρακτικές από τις ε, κοινότητες, όνομα, τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε και να τα μεταφέρουμε και σε άλλες κοινότητες. Μπορούμε να εστιάσουμε περισσότερο και στη συζήτηση που θα έχουμε με τους σκιώδεις ηγητές. Υπάρχει ακόμα πολλοί χώρους να προσθεθούν και άλλα στην έκθεση όπως έχει σήμερα. Απαντώ λίγο στον κύριο Βανίστερόι, αν θέλετε να πω ονόματα και διευθύνσεις, name and shame, να κατονομάσουμε κάποιους και να τους διαπομπεύσουμε. Η ίδια μου χώρα, η Γερμανία. Χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να καταλάβουν οι κοινότητες ότι χρειάζεται στρατηγική για τους Ρωμά. Ε, ε, για, τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Και το ίδιο ήταν, ε, σε αυτά που είπε η κυρία Γκίφεϊ, έχει αλλάξει νοοτροπία, αλλά χρειάστηκε χρόνος. Πριν από δύο χρόνια ακόμα δεν ήταν τέτοια η προσέγγιση. Σταματώ εδώ και σε αυτό το πνεύμα να δώσουμε θετικά κίνητρα, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να ε, λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και αρχίζω από την ίδια μου τη χώρα. Το πρόβλημα της υποπορόφηση είναι γεγονός. Υπάρχουν τα κονδύλια και τα κράτη-μέλη δεν τα δαπανούν, δεν τα χρησιμοποιούν. Θα πρέπει να δούμε τα διάφορα χρηματοδοτικά ε, σχήματα που υπάρχουν. Αλλά και εδώ το νόμισμα έχει δύο όψεις γιατί από τη μια έχουμε την δημιουργία δυνατοτήτων και την έλλειψη ε, γνώσης πολλές φορές, την απειρία των ίδιων των κοινοτήτων που είναι πρόβλημα. Αν θέλουμε έχουμε μια θετική προσέγγιση μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ένα τελευταίο. Ναι, γνωμοδοτεί η Επιτροπή Απασχόλησης και γίνεται μεγάλη αναφορά στην ε, μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας αλλά και σε άλλα θέματα. Και ε, τη συμπεριλαμβάνει και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες. Να δούμε πώς θα συμπεριλάβουμε τη γνωμοδότηση αυτή. Και ένα τελευταίο, τελευταίο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σημείο 3. Περίμενα να το σχολιάσετε. Αναφερόμαστε σε μια γραπτή ερώτηση που είχαμε απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε να σας πούμε ως feedback ότι μας απαντήσατε και για τα χρήματα ε, που δαπανήθηκαν μετά ε, την τροποποίηση του κανονισμού το 2010. Ήταν πολύ ανεπαρκής η απάντηση. Μήπως θα μπορούσατε να ενημερώσετε καλύτερα για το πώς απορροφήθηκαν αυτά τα χρήματα. Θα μας βοηθούσε να βελτιώσουμε και την έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι και σας προσκαλώ όλους στο ε, γεύμα που θα έχουμε για τη δικτύωση. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα καταληκτικά σχόλια για τη σημερινή μας ακρόαση και θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Στην ημερήσια διάταξη και με πολύ μεγάλη χαρά σας ενημερώνω ότι έχουμε τον κύριο Τζοβάνι Κέσλερ ενώπιόν μας. Ήδη έχει φτάσει. Περιμένουμε να μπει στην αίθουσα. Just to, to remind you that the cohesion policy... Θυμίζω ότι η πολιτική συνοχής απορροφά το 1 τρίτο του κοινοτικού προϋπολογισμού, άρα είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι τα δημόσια ε, χρήματα, που τελικά είναι χρήματα των φορολογουμένων, δαπανώνται με το σωστό και με σόφρονα τρόπο. Ε, και πάλι... Όμως μετά από τις περικοπές στον προπολογισμό και τις ανάγκες για οικονομίε σε πολλά κράτη-μέλη έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία να ε, υλοποιείται και να εκτελείται όσο γίνεται καλύτερα ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός και οι παρατυπίες και οι απάτες να περιορίζονται στο ελάχιστο ή δυνατό. Uh, ε, έλεγα λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να δαπανώνται σωστά τα κονδύλια με ένα χρηστό τρόπο. Ε, εισαγωγικά κάθε χρόνο η δυνατο ελεγα λοιπον ποσο σημαντικο ειναι να δαπανωνται σωστα τα κονδυλια με ενα χρηστο τροπο εισαγωγικα καθε χρονο η ολαφ εκδίδει έκθεση για τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητε της στο παρελθόν έτος πολλές πολιτικές ομάδες ζήτησα να προσκαλέσουμε τον κύριο Κέσλερ, όπως και έκανα, στη σημερινή συνεδρίαση για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο που θα προχωρήσουμε στο μέλλον στην πολιτική συνοχή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέσλερ για μια σύντομη παρουσίαση, ένα τέταρτο περίπου σας φτάνει και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής για σχόλια και ερωτήσεις αρχής γενομένης από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Έχετε το λόγο κύριε Κέσλερ. Um, thank you for the invitation. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω κάπως το έργο της ΟΛΑΦ. Θα επικεντρωθώ όμως ε, κυρίως σε θέματα δικών σας αρμοδιοτήτων, δηλαδή τις απάτες που διαπράττονται εις βάρος των διαρθρωτικών ταμείων. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, Υποβάλαμε την ετήσια μας έκθεση πριν από λίγες εβδομάδες και χθες την παρουσιάσαμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται να έχω μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας. Πρώτη αλλά όχι τελευταία σίγουρα. Ευελπιστώ ότι θα είναι η απαρχή μιας πολύ καλής συνήθειας που θα αξιοποιήσουμε όλοι. Ξεκινούμε με την πρώτη διαφάνεια και κάποιες γενικές παρατηρήσεις με βάση τις έρευνές μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουμε και φαίνεται και από τα νούμερα βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ιδιαίτερα στον τομέα των διαφορετικών δαμείων, έχουν όλο και μεγαλύτερη ενημέρωση, εγρήγορση και ε, αυξημένες προσδοκίες από τις αρμόδιες αρχές ότι θα αντιδράσουν πατάσσοντας τη διαφθορά και την απάτης ό,τι αφορά τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Είστε αιρετοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, είστε ευρωβουλευτές, οπότε γνωρίζετε καλύτερα από μένα πόσο επαγρυπνούν και όλο και πιο ευαισθητοποιημένοι είναι οι πολίτες για τα θέματα αυτά. Το διαπιστώνουμε και εμείς αυτή την αυξημένη επαγρύπνηση, γιατί έχουμε όλο και περισσότερες καταγγελίες από πολίτες για κρούσματα διαφθοράς ή απάτης ε, εις βάρος των κοινοτικών ταμείων. Και, και εσείς ε, οι ευρωβουλευτές ε, πολλές φορές αποτείνεστε στην ΟΛΑΦ και μας ζητάτε να αναλάβουμε δράση. Γιατί θεωρείτε ότι οι εθνικές σας αρχές πολλές φορές δεν είναι είτε πρόθυμες είτε ικανές να αναλάβουν δράση. Φυσικά οι δικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες. Πάντως το βασικό μήνυμα είναι ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ε, και της, της κοινή γνώμη ε, σε όλα τα κρατημέλη και άρα και αυξημένε είναι οι δικές μας οι ευθύνε να αναλάβουμε δράση. Επίσης ε, διαπιστώνουμε αύξηση της τάσης ε, ε, να, γίνονται όλο και, να αποκτούν όλο και πιο διασυνοριακό χαρακτήρα αυτά τα κρούσματα απάτης και διαφθοράς. Και ακόμη και οι απλούστερες μορφές απάτης, υπερτιμολόγηση για παράδειγμα, ε, προκειμένου να αποσπαστούν περισσότερα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία, πολύ συχνά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις ε, ε, είναι σε, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μια χώρες. Ε, αυτά ακόμη και για τις απλές απάτες ισχύουν. Φανταστείτε τις περίπλοκες απάτες που εξορισμού εμπλέκουν πολύ, πολύ περισσότερες χώρες προκειμένου να αποκριθούν τέτοια παραδείγματα. Οπότε έχουμε εμπλοκή εδώ πολλών δικαιοδοσιών και ακόμη και αν τα κονδύλια χορηγούνται στην ε, Ιταλία ή την Αυστρία και εμείς στις στατιστικές μας ε, ε, βλέπουμε ότι πρόκειται για αυστριακή ή ιταλική απάτη, αλλά μπορεί ο επιχειρηματίας να ήταν ε, Γερμανός ή Γάλλος. Η ιταλικη απατη αλλα μπορει ο να ηταν γερμανος η γαλλος η τραπεζα που χρησιμοποιήθηκε για να συγκαλυφθούν τα έσοδα να βρίσκονται στην Κύπρο ή στη Δανία. Θα πρέπει λοιπόν να, να αντιμετωπίσουμε και τέτοιου είδους διασυνοριακής ή διακρατικής απάτης Κυρίως όμως ε, να την αντιμετωπίσουμε με εθνικά εργαλεία και με εθνικές αστυνομικές δυνάμεις και εθνικές δυνάμεις επιβολής ε, του νόμου. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί κάποιους περιορισμούς. Έχουμε βέβαια την ΟΛΑΦ που έχει ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και αυτό είναι ένα απλό ανέκτημα, Αλλά υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο έντονα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό και η πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αγγελική Αρχής ακολουθεί αυτή την άγουσα. Έχουμε λίγε διαφάνειες τώρα για τις δραστηριότητες τη ΟΛΑΦ, τις ερευνητικές δραστηριότητες τη ΟΛΑΦ, το κάτω τμήμα της Στήλη το γαλάζιο, δείχνει την ε, σταθερή τάση των καταγγελιών που λαμβάνουμε από το 2010 είχαμε λιγότερο από 1.000 καταγγελίες. Πέρυσι το 2014 είχαμε 1.400 ε, καταγγελίες. Φέτος ήδη έχουμε 1.500. Οπότε έχουμε μια ανωδική, ε, ανωδική πορεία του αριθμού των καταγγελιών. Και αυτή είναι μια μόνιμη τάση. Τα τελευταία τρία χρόνια μάλιστα είδατε ότι αυξήθηκαν το 80% οι έρευνες που ξεκινούμε και οι έρευνες που κλείνουμε. Πέρυσι ήταν 250 οι έρευνες που έκλεισαν και ο αριθμός των συστάσεων που εκδίδει η ΟΛΑΦ, γιατί ε, κατά το πέρας της έρευνας η ΟΛΑΦ ε, ε, δίνει συστάσεις που είναι επιθαρχικού, χρηματοοικονομικού ή δικαιικού χαρακτήρα, δικαιοδοτικού. Πέρυσι είχαμε ρεκόρ συστάσεων, 400 περίπου. Και μάλιστα αυτό ήταν το ρεκόρ μας ε, πέρυσι σε ό,τι αφορά το άνοιγμα, το κλείσιμο ερευνών και την έκδοση συστάσεων. Φέτος <laughs> και μάλιστα ε, φέτο έχουμε ακόμη και λιγότερου πόρου, αλλά οι πόροι μα δεν έχουν αλλάξει οι ανθρώπινοι πόροι τα τελευταία δέκα χρόνια. Με το ίδιο προσωπικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αυξημένο εργασιακό φόρτο. Τώρα, κάτι που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Βλέπετε μια κατανομή των ε, πληροφοριών που λαμβάνουμε είτε από ιδιωτικές ή από δημόσιες πηγές. Ε, πέρυσι είχαμε 1.300 περίπου καταγγελίες, 550 από αυτές 549 για την ακρίβεια, αφορούσαν τα διαρθρωτικά ταμεία. Το 1 τρίτο, πάνω από το 1 τρίτο. Τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο το κοινωνικό. Σημαντικό λοιπόν και έρχεται σε πύρωση των αρχικών μου σχολείων. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Κάτι που φαντάζομαι θα σας κινήσει το ενδιαφέρον και Μπορούμε να σας στείλουμε τις διαφάνειες αυτές. Μερικές υπάρχουν και στην έκθεση, μερικές όμως διαφάνειες έγιναν ε, ειδικά για σας σήμερα. Θα σας τις στείλουμε μετά το πέρας της συνεδρίασης, αν ενδιαφέρεστε. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη διαφάνεια δεν υπάρχει στην έκθεση, στην ετήσια έκθεση. Κάνω λάθος? Όχι, αυτή έγινε η διαφάνεια ειδικά για σας σήμερα. Και Φυσικά χρειάζεται χρόνο για να διαβάσετε ολόκληρο τον πίνακα. Ναι, ναι, θα τις μοιράσουμε τις διαφάνειες μετά το πέρα σα για να έχετε την ευκαιρία να τις εξετάσετε πιο διεξοδικά. Εδώ έχουμε μία κατανομή των πληροφοριών που λάβαμε και έχουμε λάβει 449 πληροφορίες και καταγγελίες για τα διαρθρωτικά ταμεία. Και βλέπουμε την κατανομή ανακράτως μέλος αυτών των καταγγελιών. Και επίσης ε, το διαχωρισμό μεταξύ των ε, δημόσιων πηγών που είναι οι δημόσιες αρχές και των ε, ιδιωτικών πηγών που είναι οι πολίτες. Έχουμε αποκλείσει από τον πίνακα τις ανώνυμες καταγγελίες, γιατί από τη στιγμή που είναι ανώνυμες δεν μπορούμε να τις κατατάξουμε σε καμία χώρα. Σε μερικές χώρες έχουμε ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες, είτε από τις δημόσιες αρχές, αλλά έχουμε πολλές καταγγελίες από τους πολίτες. Ένα τέτοιο φαινόμενο ε, σηματοδοτεί ένα, πρόγραμμα, ένα πρόβλημα για το συγκεκριμένο κράτος μέλος, όταν οι πληροφορίες προέρχονται μόνο από τους πολίτες. Όταν έχουμε πολλές κατηγορίες από, και καταγγελίες από τις δημόσιες αρχές, αυτό είναι καλό σημάδι για μας, που δείχνει την ετοιμότητα των δημοσίων αρχών να πατάξουν διαφθορά και απάτη. Βέβαια αυτή είναι η δική μας ερμηνεία, μπορείτε να υιοθετήσετε κάποια διαφορετική ερμηνεία. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, την έβδομη. Εδώ έχουμε μια κατανομή των ε, τρεχουσών ερευνών της ΟΛΑΦ. Είναι περίπου 500 αυτές που διεξάγονται από πέρυσι ε, τις 31 του μηνός, 31 Δεκάτου. Ε, μεγαλύτερος ε, αριθμός αυτών των ε, ερευνών, το 1 τρίτο τους, αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία. Δηλαδή καταγγελίες απάτης και διαφθοράς που σχετίζεται με τα διαρθρωτικά ταμεία. Επόμενη διαφάνεια. Μία κατανομή ανά κράτος, μέλος. Ούτε και αυτή η διαφάνεια υπάρχει στην έκθεση. Γιατί επικεντρώνεται στα διαρθρωτικά ταμεία για το κοινωνικό και έγινε για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Η διαφάνεια αυτή, ο πίνακα αυτό σα δίνει μια ακριβή ιδέα για τον αριθμό των ερευνών που γινόνται για τη χρήση διαρθρωτικών ταμείων και που ολοκληρώθηκαν το 2014. Η κατανομή γίνεται ένα κράτο μέλος. Για το πώς έγινε η έρευνα στο κράτος και γίνεται με βάση το κράτος που διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα κονδύλια. Όπως είπα όμως η απάτη μπορεί να είναι διασυνοριακή. Βλέπετε ε, το Βέλγιο πρώτα. Μπορεί η, η μία αυτή έρευνα που ολοκληρώθηκε να αφορούσε βουλγαρική επιχείρηση. Η πορτογαλική εταιρεία. Ή να εμπλέκονται περισσότερες χώρες στην έρευνα. Αλλά πιστώθηκε το πέρας της έρευνας στη χώρα, εμπροκειμένου το Βέλγιο, που ε, απορρόφησε και διαχειρίστηκε τα διαρθρωτικά κονδύλια. Εδώ βλέπετε τα ποσά που έχει προτείνει για ανάκτηση η ΟΛΑΦ για τα διαρθρωτικά ταμεία μόνο. Στην περσινή μας έκθεση ζητήσαμε να ανακτηθεί το ρεκόρ 900 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πραγματικά ποσό ρεκόρ για την ανάκτηση και αφορά όλες τις δραστηριότητες ΟΛΑΦ. 475 εκατομμύρια, πάνω από το μισό λοιπόν των συστάσεων για ανάκτηση, αφορούσε τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό είναι το ποσό που συστήσει η ΟΛΑΦ να ανακτηθεί. Και έχουμε την κατανομή αναχώρα. Επαναλαμβάνω, σπάσαμε το ρεκόρ φέτος. Και υπάρχουν διακοιμάνσεις από χρόνια σε χρονιά. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε τάσεις γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Έχουμε αύξηση των ερευνών και αύξηση των συστάσεων και σε τελική ανάλυση αυξάνεται και το ποσό που συστήνουμε προς ανάκτηση. Μερικές έρευνες αφορούν μόνο 20.000 ευρώ, ας πούμε. Άλλες αυτή που βλέπετε στην Ισπανία και μία έρευνα αφορούσε πάνω από 200 εκατομμύρια για ανάκτηση. Εμείς προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στα μεγαλύτερα ποσά. Πάντως γενικώ είναι σημαντικά τα ποσά και παραλαμβάνω φτάσαμε σε ρεκόρ το 2014. Συνεχίζουμε. Εδώ βλέπετε τα ποσά που έχουν όντως ανακτηθεί πέρυσι από τις ε, αρμόδιες αρχές, οικονομικές αρχές, δημοσιονομικές αρχές. Μερικές φορές η ανάκτηση από τις αρμόδιες δημοσιονομικές αρχές είναι πολύ χρονοβόρα, μπορεί να κρατήσει χρόνια ολόκληρα ή να μην γίνει ποτέ, επειδή μια συγκεκριμένη επιχείρηση χρεοκόπησε για παράδειγμα. Πάντως είναι χρονοβόρα σε κάθε περίπτωση η ανάκτηση και μπορεί να γίνει είτε με δόσεις ε, και στο τέλος της δημοσιονομικής χρήσης αρχίζει η ανάκτηση ή μπορεί να αρχίσει μετά από μία πενταετία. Οπότε είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα η διαδικασία. Και η τελευταία μου διαφάνεια, γιατί έχω εξατλήσει και το χρόνο μου, ναι. και πάλι έγινε αποκλειστικά για σας, ειδικά για τη σημερινή συνεδρίαση, η σχετική διαφάνεια. Ο τίτλος είναι κάπως αποκρυφιστικός. Θα σας τον αποκρυπτογραφήσω λοιπόν. Η διαφάνεια αυτή ε, συγκεντρώνει ανά χρόνο τις ατασταλίες και τις απάτες που έχουν ε, ε, ανακαλυφθεί από τα κράτη-μέλη ατασταλίες και απάτες που έχουν ανακαλυφθεί από τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη οφείλουν να, να ενημερώνουν, να υποβάλουν έκθεση για τέτοιου είδους ατασταλίες και απάτες. Και έχουμε και τα ποσά που ε, προτείνει η Όλαφ για τις ανακτήσεις. 475 ε, ε, είχαμε και το 2014 πρόταση για ανάκτηση ποσών. Η γαλάζια στήλη είναι ε, οι αποκαλύψεις που έκαναν τα κράτη-μέλη για τις ατασταλίες, οι αναφορές που έκαναν για τις ε, ατασταλίες που ανακάλυψαν και η δεύτερη τελευταία στήλη είναι τα ποσά που εμείς προτείναμε για ανάκτηση. 45 ερευνητές ε, ασχολούνται ιδιαίτερα με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα γεωργικό ταμείο. Μόνο με αυτά. Έχουμε 45 και το 2002. 2,5% του συνόλου των ατασταλιών που αποκαλύφθηκαν έγιναν από τους 45 ε, ερευνητές. Το 2013 ήταν 8% και το 2014 ήταν 25%. Κάνουμε πολύ σοβαρό αργό και μάλιστα μερικές φορές ε, δυσανασχετούν τα κρατημέλη γιατί όταν λαμβάνουν σύσταση από εμά για ανάκτηση 200 εκατομμυρίων ε, δεν πετάνε και από τη χαρά τους. Αλλά βλέπετε τι αντίκτυπο έχει το έργο μας ε, στα κρατημέλη και τι αλληλεπίδραση έχουμε. Ελπίζω να σας έδωσα έστω και μια επιφανειακή ε, ιδέα για το ποιο είναι το έργο της ΟΛΑΦ και σας έδωσα και κάποια τροφή, αριθμούς είναι συγκεκριμένα, για σκέψη και για περαιτέρω συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και ευχαριστώ που ετοιμάσατε και ειδικέ διαφάνειες και ειδική ενημέρωση για την Επιτροπή μας. Θα μοιράσουμε τις σχετικές πληροφορίες. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής που το επιθυμούν. Και ξεκινώ με τους συντονιστές, ο κ. Βανίστελ Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θαυμάσιο αυτό έγγραφο. Την έκθεση είναι και πολύ χρωμή. Έχω μερικές ερωτήσεις για τα διορθωτικά ταμεία και κάποιες γενικές συζητήσεις βέβαια που θα ακολουθήσουν θα είναι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολογισμού όπου εκεί είστε συχνός επισκέπτης και προσκεκλημένος μας. Ε, γενικές ερωτήσεις λοιπόν. Εδώ βλέπω στην ενημέρωσή σας ότι είναι αρκετά γενικόλογοι. Και τώρα βλέπω ότι υπάρχουν τρεις χώρες. Η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ισπανία που εστιάζεται, όπου εστιάζεται μάλλον ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό έχει σημασία. Θέλω να δω την κατανομή ε, στην ε, τακτική σας έκθεση. Όχι, όχι, για την Όλαφ. Πολλά λέτε, εντάξει, αλλά λιγότερα λέτε για το πώς κατανέμεται αυτό αναχώρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ίσως στο μέλλον να το σκεφτείτε αυτό. Ήδη στην έκθεσή σας να αναφέρονται τα κράτη-μέλη. Και να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή να σας τη δώσει. Αλλιώς πώς θα δουλέψουμε εμείς. Γιατί δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω κάθε φορά. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Τώρα που έχετε αυτά τα στοιχεία που είναι και ψηλά. Ε, είναι πρόσφατα. Δηλαδή από πότε τα έχετε. Σε ποιες εποχές αναφέρονται. Το 2004. Πού ανάγονται. Στο 2013. Είναι παλιές περιπτώσεις. Από πότε έχουν συσσωρευτεί αυτές. Ποιο έτος αφορούν, την παλιά περίοδο, τη σημερινή. Είναι υποθέσεις ετών που διονίζονται. Ή μπορούμε να πούμε εντάξει, αλλάξαμε τους κανονισμούς μας, μας γίναμε πάρα πολύ σκληροί για τους ελέγχους, για το αποτέλεσμα και κάναμε και πάρα πολλές άλλες αλλαγές. Ε, στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Επιτροπή μας Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ρέτζη. Λοιπόν, αυτές όλες οι υποθέσεις που συσσωρεύονται είναι σημερινές, χτεσινές ή προχτεσινές και προπέρσινες. Ε, θέλω να ξέρω σε ποια περίοδο αναφερόμαστε. Και για τα υπόλοιπα, καμιά φορά έχω ενημέρωση από άλλα κρατημέλη και πάμε αμέσως στην Όλαφ και λέμε ορίστε, έχω αυτή την ενημέρωση, τι να την κάνω. και ξέρω ότι η αντιμετώπιση συχνά ήταν οργισμένη. Έρχεται ένας δημόσιος υπάλληλος, σας τα λέει, ε, σας δίνει χαρτιά, τα παίρνετε, τα, ε, κινείται κάποια διαδικασία και η έκβαση είναι δική σας ευθύνη. Αλλά έρχονται και στους ευρωβουλευτές και τα λένε αυτά και δεν ξέρουμε τι συνέχεια δίδεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ ο κύριος Βον, εξ Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και χθε ο κύριο Κέσλε ήρθε στην Επιτροπή αυτή με την ετήσια έκθεσή του και νομίζω ότι πολλά μέλη ικανοποιήθηκαν από τις βελτιώσεις στα νούμερα που μας παρουσίασε ο κύριο Κέσλερ. Βεβαίω, τέθησαν πολλέ ερωτήσει ε, χθες. Κάτι ακόμα που ήθελα να τονίσω όταν μιλάω για αυτό το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ε, τη και την απάτη και το ποσοστό σφάλματος και την απάτη. Ορισμένοι λένε ότι μόλις πούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, αμέσως λένε και πω από τι τεράστιο ποσοστό είναι αυτό. Το ποσοστό απάτης είναι πολύ χαμηλό, είναι γύρω στο 2% και πολλά κράτη-μέλη θα ήθελαν να έχουν χαμηλό, ε, τόσο χαμηλό ποσοστό στις απάτες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα και γι' αυτό και ο κύριος Κέσλερ ήρθε χθε στην Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού και σήμερα εδώ. Ε, και είναι πολύ σημαντικές οι παρουσιάσεις του. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι οι διαφορές στα κράτη-μέλη σε σχέση με τις υποθέσεις που αναφέρονται, που ερευνώνται και που ολοκληρώνονται και αυτές στις οποίες έχουν υπάρξει ε, καταγγελίες, ε, ένα σωρό πολλές φορές, ε, υπάρχουν μάλλον ένα σωρό υποθέσεις όπου τα νούμερα δεν αντιστοιχούν ε, υπάρχουν δηλαδή κάποια σύγχυση. Η πρώτη μου ερώτηση είναι τι πιστεύει, σε τι πιστεύει ότι οφείλεται αυτό ο κύριος Κέσλερ, επειδή το κάτω μέλος έχει διαφορετικό σύστημα αναφοράς της απάτης, έρευνας της απάτης ε, και αν ναι, όπως φαντάζομαι ότι ισχύει, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, ώστε να έχουμε ε, συγκρίσιμα και συνεπίστοιχες ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ε, ε, σε 475 εκατομμύρια για τα διευθυντικά ταμεία, ποσοστό, μάλλον χρήματα τα οποία είναι ανάκτηση. Όταν μιλάτε λοιπόν για αυτά τα, την κάλυψη αυτών των χρημάτων, ξέρετε τελικά πόσα όντως ανακτώνται μετά από τις δικές σας συστάσεις. και αυτό είναι το, το βασικό ζήτημα. Όταν δούμε επίσης τα υπόλοιπα στοιχεία, ε, ε, με εντυπωσιάζει πόσο χαμηλό είναι το προσωπικό. Έχετε πρόβλημα στη στελέχωση. Ε, ε εσείς ε, πρέπει να κάνετε 5% περικοπές στο προσωπικό όπως όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και είναι πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάνα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και για την έκθεσή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, Είπατε ότι το μισό ποσό ανακτήσεων που συνιστάται είναι από τα διαρθωτικα ταμεία. 475 76 ε, εκατομμύρια είναι πολύ ψηλό από τα διαρθωτικά ταμεία. Το επόμενο είναι αναπτυξιακή βοήθεια που είναι 174. Και είπατε ότι είναι ελάχιστα τα ποσά που έχουν ανακτηθεί. 22 νομίζω, κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πολύ απλή. Ποια είναι η πρακτική και η πολιτική συνέχεια που δίδεται με αλφαγιώτα σε μια τέτοια έκθεση. Πάρα πολλέ συστάσει απευθύνεται εσεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα κράτη-μέλη. Εκείνοι ε, τι εφαρμόζουν, συμμορφούνται και αν όχι, τι συμβαίνει. Μπορείτε να μα δώσετε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα έρευνας και στα διαρθρωτικά ταμεία ας πούμε και τι συνέχεια δίνεται και τι έκβαση τελικά ε, επιτυχάνεται. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση είναι της κυρίας Δαμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κέσλερ, τον Διευθυντή, για την ενημέρωση και τα στοιχεία που μας έδωσε. Τα διευθυντικά ταμεία είναι οικονομική συμβολή. Είναι ένας από τους τομείς από τους οποίους έχουμε τις περισσότερες πληροφορίες και επί του οποίου φυσιολογικά επικεντρώνεται η προσοχή της όλα. Συμφωνώ μαζί σας ότι με υψηλότερο ε, ε, αριθμό καταγγελιών δεν σημαίνει απαραίτητο περισσότερες απάτες. Όμως δείχνει περισσότερη ενεργητικότητα από πλευρά της διοίκησης και των πολιτών. Σας ρωτώ λοιπόν από τα όσα είδατε, κυρίως ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά πίσω από τις απάτες στον προπολογισμό της Ένωσης κρύβονται συμφέροντα του, εγκληματικού, του οργανωμένου εγκλήματο. Υπάρχουν μηχανισμοί κατά τη γνώμη σας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά πέρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από πλευρά τη διοίκηση των κρατών μελών, αλλά και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μπορούσαν να παρεύουν, α πούμε η σύσταση ειδικών επιτροπών, οι ομάδε εργασία. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι δεσμευμένη και για το θέμα του περιβάλλοντο δεδομένη τη γεωγραφική μου προέλευση, έχουμε σημειώσει ιδιαιτερότητε μάλλον κακή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που συνδέονται με περιβαλλοντικά εγκλήματα. Να χρησιμοποιούνται δηλαδή υποτίθεται τα ευρωπαϊκά χρήματα για να σταματήσουν περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά τα χρήματα καταλήγουν στα λάθος χέρια χωρίς να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Και η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και από δικής μου πλευράς, κύριε Διευθυντά, για αυτή την εισήγηση που θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να μελετήσουμε καλύτερα στη συνέχεια. Μια ερώτηση κάθετος παρατήρηση σε σχέση με τα νούμερα που μας δώσατε. Φαίνεται να υπάρχει μια πορεία, όπως είπατε, τυχαία. random όπως είπατε, αλλά σίγουρα με αύξηση της σύστασης ε, ανακτήσεων ε, κονδυλίων μέσα στο 2014 και ίσως ε, αυτό αν μπορούσε κανείς να κάνει μια σύγκριση θα βλέπει και αύξηση, μια τάση για αύξηση καθώς περνούν τα χρόνια. Τα χρόνια κυμαίνονται βέβαια γιατί η έρευνα δεν διαρκεί πάντα, ίσως να διαρκεί ένα χρόνο. Δηλαδή από τον ένα χρόνο στον άλλο να γίνονται έρευνες που δεν επιτρέπουν να πούμε ότι σε εκείνο, τη φάση, σε εκείνο το χρόνο αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβω είναι η εντύπωσή σας πέρα από τα νούμερα που θελω να καταλαβω ειναι η εντυπωση σας περα απο το νουμερα που ενταξει μας λένε κάποια πράγματα, η εντύπωσή σας είναι λοιπόν ότι η, η αύξηση των ε, χρημάτων που πρέπει να ανακτηθούν οφείλεται σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της Όλαφ και καλύτερη συνεργασία με τα κράτη ή συνδέεται με επιδίνωση στη χρήση των κονδυλίων. ίσως με την κρίση να υπάρχει μια αύξηση της τάσης για απάτες. Είναι τυχαίο, γιατί εντάξει υπάρχει μια ισπανική υπόθεση μεγάλων διαστάσεων που ίσως να άλλαξε να, τα, τα νούμερα. Θέλω να καταλάβω λοιπόν ποια είναι η εντύπωση δική σας για τα νούμερα, για να καταλάβω αν πρέπει να ανησυχούμε. ή ε, όχι, αν θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι αντίθετα, γιατί εν γέννη επιτυχάνεται καλύτερα ο στόχος της αποφύγης των απατών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Είχα την ίδια ερώτηση με την ε, συνάδελφο Βάνα. Δηλαδή, τι γίνεται με την ανάκτηση γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό της ανάκτησης ε, που προτείνει η ΟΛΑΦ από τα κράτη-μέλη. Και έχω και μια άλλη ερώτηση. Ποια η διαφορά ατασταλίας και απάτης. Τη στιγμή που δεν υπάρχει δόλος, ε, αλλά απλώς ατασταλία τι γίνεται, ή σε περίπτωση που νομίζετε ότι αρχικά δεν υπάρχει δόλος, αλλά στην πορεία διαπιστώνεται ότι Είσαι ατασταλία είχε γίνει τελικά εσκεμμένα, άρα υπάρχει απάτη. Επίσης, τι επαφή έχετε με τις περιφερειακές αρχές, γιατί οι περιφέρειες είναι πολλές φορές δικαιούχοι των διαρθρωτικών ταμείων και διαρθρωτικών κονδύλιων. Έχετε επαφή μαζί τους, επικοινωνείτε μαζί τους και πώς. Στην Τσεχία, εκκρεμωδική μία υπόθεση όπου ένας περιφερειάρχης δωροδοκούντο, χρηματίζονται και μάλιστα ε, συνελήφθη επαυτοφόρο να λαμβάνει ε, φακελάκι ε, σε ένα μπουκάλι κρασί, μέσα σε ένα μπουκάλι κρασί. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν τέτοιου είδους ε, προσεγγίσεις. Ο κύριος να ευχαριστώ. Κύριε Γενική Διευθυντά μου, καταρχάς πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη να έχουμε ενιαία ερμηνεία των νόμων για ε, τις δημόσιες συμβάσεις που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλιώς έχουμε εθνικές αναγνώσεις, εθνικές ερμηνείες και προβλήματα που απορρέουν από την ερμηνεία στις Βρυξέλλες. Τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, το είπαν και οι συνάδελφοι. Υπάρχει σαφής ανάγκη να ξεκαθαριστεί η νομική συμπεριφορά και, και, μοίρα που επιφυλάσσουμε στις δύο κατηγορίες, τα σφάλματα και τις απάτες. Από νωρίς, από αρχικό στάδιο θα πρέπει να γίνεται αυτό και να έχουν τις ίδιες συνέπειες γιατί οι καθυστερήσεις ή ε, ε αναστολή της χρηματοδότησης μέχρι να ξεκαθαριστεί, αυτό οδήγησε σε τεράστια προβλήματα με τεράστιες καθυστερήσεις που έχουν δύο βασικούς χαμένους ε, τους ε, ενδιαφερομένους, τις κοινότητες και τους συμβασιούχους. Ε, δεν μπορείς να περιμένεις έξι μήνες και ένα χρόνο να μην έρχονται τα χρήματά σου και μετά από έρευνα ενός έτους να σου λένε ότι όλα εντάξει είμαστε μια χαρά αλλά έχεις πεθάνει Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Είτε θα επιταχύνουμε τη διαδικασία, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον, είτε θα έχουμε δύο διαφορετικά νομικά ε, φάρμακα εντό εισαγωγικών, γιατί άλλο πράγμα είναι το σφάλμα και άλλο πράγμα είναι η απάτη. Έρχομαι τώρα σε ένα περιστατικό από τη Ρουμανία, γιατί επί σειρά ετών η Ρουμανία, όχι μόνο, αλλά κυρίως η χώρα μου, ήταν μια περίπτωση μελέτης. Το 2011, τον Ιούνιο, υπήρξε ένα εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέφερε ε, τη συνεισφορά της Όλαφ. Και εγώ θα προσπαθήσω τώρα να το παραθέσω όσο το θυμάμαι, με όση ακρίβεια. Θεωρεί λοιπόν η Όλαφ ότι συντονίζονται διάφορα υπουργεία ε, στη Ρουμανία για να αντικρούσουν και να εμποδίσουν την έρευνα της Όλαφ. Κάπως έτσι το έλεγε αυτό το έγγραφο, του οποίου είχε γνώση ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι ε, αξιωματούχοι και υπάλληλοι. Ε, μόλις τον Οκτώβριο του 2012 όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει Έξι, έξι μόνο λειτουργικά προγράμματα επιχειρησιακά με πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για μήνες ολόκληρους. Λύθηκε μεν το πρόβλημα, αλλά η Ρουμανία σήμερα αντιμετωπίζει τεράστια πίεση για να απορροφήσει στο υπόλοιπο διάστημα αυτά τα τεράστια χρήματα, διότι υπάρχει δυσκολία ε, και μόνο να διοχετευτούν στο τραπεζικό σύστημα για να πληρωθούν οι παραχωρησιούχοι, οι συμβασιούχοι. Αυτή η καθυστέρηση εχει τεράστια ολέθρια αποτελέσματα. Θα πρέπει σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχει ένα πρόβλημα να αποφασίζετε εσείς να το σταματήσετε. Α, το σταματάτε ένα χρόνο μετά με όλα τα συμπαρομαρτούντα δεν είναι μόνο άδικο, είναι και επικίνδυνο και αντίθετο με την ίδια την πολιτική ε, συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρο. Ο κύριος Ραπέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση και η έκθεση πολύ χρήσιμη γιατί μας επιτρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα την κατάσταση και να εξετάσουμε, να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των διαφόρων χωρών. Εσείς ε, αναλύετε τις καταγγελίες, ε, πραγματοποιείτε έρευνες και προσπαθείτε να εντοπίσετε απάτες ή ατασταλίες. Έχουμε όμως ε, περιπτώσεις τεράστιων προγραμμάτων. Προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε με διαφάνεια αλλά διαπιστώνουμε τελικά ότι κατασπαλήθηκαν κονδύλια εξαιτία ε, τη αναποτελεσματική χρήση των κονδύλιων. Πέραν το απάτη, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην αποτελεσματικότητα τη διαχείριση των κονδύλιων. Αυτό το εξετάζεται και προβαίνεται τάσει ε, σε περίπτωση αναποτελεσματικής χρήσης ε, των κονδυλίων από κάποια χώρα. Οι χώρες διαφέρουν μεταξύ τους. Άλλες έχουν πιο κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Οι βαλτικές χώρες, για παράδειγμα, ε, ολόκληρη χώρα είναι μία περιφέρεια. Οπότε ο σχεδιασμός γίνεται κεντρικά και αποφασίζεται ποια συγκεκριμένη περιοχή θα επωφεληθεί και ποιο πρόγραμμα θα δρομολογηθεί. Άλλες χώρες έχουν πιο αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης. Κατά τη γνώμη σας, ε, ποια μέθοδος είναι η καλύτερη, η πιο κεντροσχεδιασμένη ή η αποκεντρωμένη οι χώρες που είναι πιο επικεντρωμένες και αφήνουν τα πράγματα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις χώρες που έχουν συγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο των προγραμμάτων. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον για να δούμε και στο μέλλον ποια είναι η καλύτερη μέθοδος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αλλά κυρία Μάλετιτς και καλώς ήρθατε κύριε Κέσλερ. Σας ευχαριστούμε και για την παρουσίαση και για τις διαφάνειες που ετοιμάσατε ειδικώ για, για μας. Πολύ ενημερωτικές και χρήσιμες. Ε, διαπιστώστε τη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών. Ε, έχουμε κράτη-μέλη που δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία για οι καταγγελίες, ε, δεν λαμβάνετε καθόλου καταγγελίες ούτε από τον δημόσιο, αλλά έχετε και ελάχιστε καταγγελίε από ιδιώτες για, για κάποια κράτη-μέλη. Πώς ε, μεριμνάτε ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός ε, των προβλημάτων στα κράτη-μέλη. Γιατί πέραν ε, του δικτύου των αρμοδίων αρχών στα κράτη-μέλη και πέραν της προσπάθειας που γίνεται στην επιμόρφωση, έχουμε και κάποιες εθνικές στρατηγικές που δίνουν έμφαση στην πρόληψη, στον εντοπισμό των ατασταλιών, αλλά και κάποιες δραστηριότητες επιμόρφωσης για αποτροπή. Αλλά είναι πραγματικά πολύ σοβαρό αν δεν έχετε καθόλου πληροφορίε ή καταγγελίε από κράτη-μέλη ούτε από το δημόσιο τομέα ούτε από τι ιδιώτε, γιατί αυτό είναι απόδειξη ότι το σύστημα στην πράξη δεν λειτουργεί. Επίση, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια αύξηση των καταγγελιών και των πληροφοριών, αλλά ταυτόχρονα μείωση του αριθμού των ερευνών που ξεκινάτε. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Ευχαριστώ κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κέσλερ για τις πληροφορίες. Έχω μερικές ερωτήσεις. Θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε σχετικά με τις δραστηριότητες της Όλαφ. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να έχεις καθήκον ε, να διαφυλάσεις το δημόσιο χρήμα. Αλλά Μαθαίνω από δημοσιεύματα ότι κάποια στιγμή υπήρχαν 423 όσεις που, έρευνας που άνοιξαν ε, την ίδια μέρα για εταιρείε κυρίως στη Βουλγαρία και την ε, Ρουμανία. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί από όσα μαθαίνουμε και είναι δημόσια αυτά τα στοιχεία. Πολλές από τις έρευνες αυτές διακόπησαν ξαφνικά και ε, εγκαταλείφθησαν, δεν ολοκληρώθησαν, αλλά αυτό έπληξε τις εταιρείε ε, που ήταν υπό διερεύνηση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ε, πρόκειται για ανθρώπους, για θεσμούς, για τοπικές αρχές που επένδυσαν ε, τα λίγα χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους και κάποια στιγμή σου λένε σταματάει χρηματοδότηση γιατί είσαι υπό έρευνα. Η έρευνα ολοκληρώνεται ή δεν ολοκληρώνεται, εγκαταλείπτεται ε, δεν αποκαλύπτει τίποτα παράνομο, ε, αλλά η χρηματοδότηση έχει χαθεί. Θα ήθελα παρακαλώ να μου απαντήσετε ρητά. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα απογίνουν. Άλλο είναι η απάτη, την οποία φυσικά και οφείλετε να πατάξετε και μάλιστα αμήλικτα, δεν διαφωνώ καθόλου, δεν χωράνε εδώ ε, παζάρια ούτε συμβιβασμοί, αλλά άλλο η απάτη και άλλο είναι το σφάλμα. Μπορεί να κάνει και ένα λάθος ένας άνθρωπος. Στη Ρουμανία, ας πούμε, η λάθος εγγραφή ας πούμε στα λογιστικά βιβλία ήταν ποσό μικρότερο των 7 ευρώ. 7 ευρώ. Δεν συμφωνούσε το ταμείο για 7 ευρώ και τους μπλόκαραν τη χρηματοδότηση. Εγώ εκτιμώ το έργο σας και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει εμπλοκή εκεί. Το συζητήσαμε και στο Στρασβούργο στην Επιτροπή μας την περασμένη εβδομάδα έχουν ε, οδηγηθεί σε εμπλοκή, τα κονδύλια δεν μπορούν να απορροφηθούν και πολλοί πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο Ρουμάνοι, αλλά και από άλλα κράτη-μέλη, έχουν αυτό το πρόβλημα και ε, διστάζουν ε, να ε, υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση, για κοινοτικά κονδύλια. Γιατί σου λένε ένα λάθος να κάνω, έχω υποθηκεύσει το μέλλον μου, την οικογένειά μου, την περιουσία μου και μπορώ να πάω και φυλακή. Οπότε καταλαβαίνετε ποιος πληρώνει αυτό το λογαριασμό, τα χρήματα που χάνονται τελικά. Ευχαριστώ. And Madame Smolkova. Κυρία Σμόλκοβα. Ευχαριστώ πολύ ε, και τον κύριο Κέσλερ για τις απαντήσεις. Αλλά η αποκάλυψη διαφόρων αξιόπινων πράξεων στα διάφορα κράτη-μέλη είναι σημαντικό. Τι γίνεται όμως τελικά με την αποκάλυψη, με τη δημοσίευση όλων αυτών και πώς προβάλλεται στον κόσμο. Αν θεωρείται αρνητικό μέτρο, ή αποτρεπτικό και ε, τι γίνεται με τα κράτη-μέλη που είναι καθαροί αποδέκτες. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι τα χρήματα αυτά είναι λεφτά που μας, μας προσφέρουν, ε, δεν είναι χρήματα του προϋπολογισμού, κάποιος μας δίνει λεφτά και ε, δεν έχουμε κανονική πρόσβαση. Ε, είναι πολύ σημαντικό να λέμε δημόσια τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Ήθελα και εγώ να θέσω μια ερώτηση ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είδα ότι υπάρχει μια ένα σύντομο κομμάτι στην ετήσια έκθεσή σας που αφορά την πρόληψη της απάτης και την ανείχνευση των ε, δραστηριοτήτων. Πώς βλέπετε το μέλλον της πρόληψης και των, της ε, απάτης και των ατασταλιών σε σχέση με το τομείο Συνοχής. Και επίσης ε, πώς θα μπορούσατε να κατατήσετε τους εθνικούς ε, φορείς. Ε? Γιατί επανειλημμένως οι συνάδελφοι ανέφεραν εδώ στην Επιτροπή ότι έχουμε προβλήματα με την ποιότητα της εργασίας των εθνικών ε, φορέων. Αυτή είναι η ερώτησή μου, ήταν και τελευταία και έχετε το λόγο, αν μπορείτε κάπως σύντομα να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Σύντομα είναι δύσκολο θα προσπαθήσω να απαντήσω γιατί όλες οι ερωτήσεις είναι σημαντικές. Και από τις δικές σας ερωτήσεις καταλαβαίνω τι θα θέλατε εμείς να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ερωτήσεις, αλλά είναι και ενδείξεις, κατευθύνσεις για μας. Θα ακολουθήσω τη σειρά με μια εξαίρεση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπούντα, γιατί ρωτήσατε επιμόνως να σας δώσω μία ε, σταθερή και σίγουρη απάντηση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Τίποτα δεν συνέβη στις εταιρείε τις οποίες ερευνήσαμε. Είναι αλήθεια ότι ανοίξαμε 219 έρευνες. Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα, ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης της ΟΛΑΦ της 1η Πρώτου 2012. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της εργασίας που είχαμε κάνει το 2011. Είχαμε κάνει δηλαδή την επιλογή ενός, μιας τεράστιας καθυστέρησης που είχαμε. Και είναι αλήθεια ότι αυτές οι έρευνες έγιναν για υποθέσεις χρηματοδότησης από τα διευθυντικά ταμεία, κυρίως στις χώρες που είναι και οι μεγαλύτεροι παραλήπτες ε, δικαιούχοι. Και σας απαντώ, αλλά απαντώ ταυτόχρονα και σε κάποιους άλλους βουλευτές. Και το λέω λοιπόν με πάσα ε, βεβαιότητα. Ε, η έναρξη μιας έρευνας της Όλαφ δεν κινητοποιεί οποιαδήποτε αναστολή χρηματοδότησης. Η έναρξη μιας έρευνας της Όλαφ δεν οδηγεί καν σε ενημέρωση των ε, χρηματοδοτικών αρχών ούτε καν για το έναρξη της έρευνας. Απλώς εμείς ξεκινάμε μια έρευνα, η οποία δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στη χρηματοδότηση. Πιθανή επίπτωση στη χρηματοδότηση προέρχεται από την πιθανή σύσταση στο τέλος της έρευνας ναι, και μόνο αν βρούμε όντως αποδείξεις. Δηλαδή η έναρξη μιας έρευνας, ούτε η ολοκλήρωση μιας έρευνας δεν οδηγούν σε καμία συνέπεια για τους ανθρώπους που είναι υποέλεγχο ή για τις εταιρείες που είναι υπό έλεγχο. Ότι η έναρξη των ερευνών δεν, οδηγεί, δεν έχει επιπτώσει. Στις 219 περιπτώσεις μάλιστα μόνο σε τέσσερι από αυτές τις υποθέσεις που ξεκινήσαμε την 1η Δευτέρου 2012 επρόκειτο για άτομα ή εταιρείε. Όλα τα άλλα αφορούσαν χρηματοδότηση. Ελπίζω αυτό να σας καθησυχάζει για το τι έγινε τότε και για το τι συμβαίνει φυσιολογικά και μάλιστα ερευνούμε ε, ε, εις βάρος ή για απαλλαγή. Δηλαδή κάποιες από τις έρευνές μας ορισμένες από τις αρκετές μάλιστα, καταλήγουν στο ότι δεν υπήρξε απάτη. Και αυτό είναι επιτυχία επίσης. Είναι πάντοτε επιτυχία όταν διαπιστώνουμε τι έγινε. Μαύρο ή άσπρο δεν έχει, δεν έχει διαφορά. Και ξεκινάμε μια έρευνα, όχι αυθαίρετα, αλλά όταν υπάρχουν ισχυρισμοί, καταγγελίες, υποψίες για απάτη. Με τη βάση σοβαρών ισχυρισμών. Και αυτό έγινε τότε και αυτό γίνεται και φυσιολογικά. Επιπλέον, στη διάρκεια μιας έρευνας μπορεί να εκδώσουμε ένα αίτημα προς την ε, Δημοσιονομική Αρχή να αναστείλει, να λάβει δηλαδή προληπτικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα όταν έχουμε σοβαρές υποψίες και συμβαίνει, δεν έχω τώρα εδώ τα νούμερα, αλλά γίνεται στο 3% των υποθέσεων. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν η έναρξη ή η διεξαγωγή μιας έρευνας ε, της ΟΛΑΦ ε, πυροδοτεί αυτό που αναφέρατε. Ελπίζω λοιπόν αυτή να ήταν ξεκάθαρη απάντηση όπως το ζητήσατε. Και τώρα θα πάμε στη σειρά. τρεις, χώρες. Υπάρχουν όλα τα... Ε, οι, προϋποθέσεις αυτές που σας είπα. Ίσως να είναι Ιταλός εργολάβος, επιχειρηματίας που έκανε τη συγκεκριμένη ε, δουλειά στη Βουλγαρία ή Γερμανός. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπόθεση στη Βουλγαρία όπου Γερμανός και Βούλγαρος επιχειρηματίας μαζί οδήγησαν σε δύο έρευνες της Όλαφ και αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν σε δύο δικαστικές ε, διώξεις, μία στη Γερμανία και μία στη Βουλγαρία. Απαντώ λοιπόν σε εσά και ταυτόχρονα και στους άλλους συναδέλφους σας που ρώτησαν ε, για τη Ρουμανία. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που έχουν ολοκληρωθεί πέρυσι. Οι περισσότερες εξ αυτών μάλιστα δεν είναι εδώ γιατί δεν είναι για τα διευθυντικά ταμεία, αλλά θα τις δείτε στην έκθεση, γιατί η έκθεση αφορά όλα τα ταμεία. Είναι υποθέσεις που αφορούν το ΣΑΠΑΤ, το προενταξιακό πρόγραμμα. Ολοκληρώσαμε. Όλες αυτές οι υποθέσεις έκλεισαν πέρυσι. Και έτσι απαντώ στην ερώτησή σας. Ε, κανονικά τα διαστατικά ταμεία και οι σχετικές έρευνες, ε, τις τελευταίες που έγιναν, αφορούν ε, μάλλον κατά μέσο όρο διαρκούν 22 μήνες. Είναι οι μακρύτερες έρευνες, οι πιο μακροχρόνιες. Κατά μέσο όρο, όταν αφορούν προσωπικό ή μέλη των θεσμών, διαρκούν 10 μήνες. Στις άμεσες δαπάνες 11 μήνες. Αυτές που αφορούν τα διευθυντικά ταμεία και την εξωτερική βοήθεια είναι οι μακρύτερες ερευνές και μπορείτε να καταλάβετε και γιατί. Γιατί πρέπει να ερευνήσουμε ε, στα κράτη-μέλη, στην κάθε περιφέρεια και, και εκτός και σε τρίτες χώρες. Οπότε εκεί χρειαζόμαστε τη συνεργασία των τοπικών αρχών της δημόσιας διοίκησης, οπότε γι' αυτό παίρνει περισσότερο χρόνο. Ναι, σύντομα, ο κύριος Αν Είναι παλιές υποθέσεις. Και οι παλιές υποθέσεις περιλαμβάνονται σε μια έκθεση ενός έτους. Και τα νούμερα ανεβαίνουν. Ας πούμε το 2014 ότι είχαμε ένα πολύ ψηλό νούμερο. Πώς επηρεάζεται από τις παλιές υποθέσεις αυτό το νούμερο και πότε κανείς μπορεί να πει ε, αμάν, χάλια πάντα πράγματα. Είναι δύσκολο να πούμε, αλλά όλες οι στατιστικές, και δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ τώρα αυτό, πρέπει να τις δούμε πώς ε, ε, σχηματίζουν, πώς δείχνουν μάλλον τις τάσεις. Είναι πιο σημαντικές οι τάσεις παρά το ετήσιο νούμερο. Αν με ρωτήσετε, και κανείς δεν μου επέβαλε άμεσα αυτή την ερώτηση, αλλά αν με ρωτήσετε, ας πούμε, ποια είναι η κατάσταση στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία είχαμε πολλές έρευνες, πολλές υποθέσεις στο παρελθόν, τις οποίες τώρα ολοκληρώσαμε, ιδιαίτερα με τα ταμεία ΣΑΠΑΡΤ, τα κονδύλια ΣΑΠΑΡΤ και υπάρχουν επίσης προβλήματα για την εφαρμογή των συστάσεών μας. Το βλέπετε σε μια άλλη διαφάνεια για τις, ε, ε, ε, την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, αλλά βλέπουμε από τα τελευταία χρόνια ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, από τότε που εγώ είμαι στην όλα τουλάχιστον. Ας πούμε, η εισαγγελία κατά της διαφθοράς έχουν λειτουργήσει εξαιρετικά, κατά την άποψή μας. Έχουμε εξαίρετη συνεργασία. Η DILAF κάνει εξαιρετική δουλειά. Εφαρμόζουν τις συστάσεις μας και κάνουμε κοινέ έρευνες ή παράλληλες έρευνες. Πραγματικά ε, είναι υπόδειγμα για τις άλλες χώρες. Και αυτό εν μέρει εξηγεί γιατί έχουμε μεγάλα νούμερα στη Ρουμανία. Συν άλλη μια εξήγηση είναι ότι οι παλιές υποθέσεις του προγράμματος ΣΑΠΑΡΤ και όλες αυτές οι υποθέσεις, αν είμαι ανοιχτό στους ευρωβουλευτές, είναι βεβαίως. Και δεν σας πιέζω, ούτε παρακαλάω για περισσότερη δουλειά. Έχω αρκετή. Αλλά αν με ρωτήσετε αν ε, τα, οι ευρωβουλευτές μπορούν να έρθουν και να αναφέρουν σε εμά πράγματα, φυσικά και μπορούν. Το κάνουν ήδη. Ήδη γίνεται αυτό και είμαστε ανοιχτοί. Δεν χρειάζεται να σας πω και δεν το κάνω μόνο για πολιτικό, το κάνω εγώ για πολιτικούς λόγους, δεν χρειάζεται να... Αυτό το έχουν κάνει κάποιοι βοηθοί, αλλά Εντάξει, γίνεται και αυτός ο τσακωμός ανάμεσα στις ομάδες. Εμάς ε, γινόμαστε αντικείμενο χειρισμών σε όλα αυτά. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και... Α, έφυγε στο μεταξύ ο κύριος Βον. Ρώτησε για τις διαφορές, τις αναφορές που κάνουν τα κράτη-μέλη. Άρα νομίζω ότι ήδη απάντησα. Και απάντησα και σε άλλη ερώτησή του που την εστερνίστηκε και μια κυρία από το κόμμα των Πρασίνων. Συγγνώμη, δεν σας ε, ξέρω, δεν σας έμαθα ακόμη. Το, ποσοστό ανάκτησης. Υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση ως προς αυτό. Όταν δείτε τη σύσταση μας μέσα σε ένα χρόνο για την ανάκτηση, 900 εκατομμύρια, και την ίδια χρονιά έχουμε ανάκτηση 200 εκατομμυρίων, είναι άσχετη η σύσταση με την ανάκτηση δεν ταιριάζουν ε, οι συστάσεις με την ανάκτηση. Ε, ο σύνδεσμος δεν υπάρχει, είναι πολύ χαλαρός. Απλώς σε ένα δεδομένο χρόνο συστήσαμε ανάκτηση 900 ε, εκατομμυρίων. Μπορεί και στις 30 Δεκεμβρίου και την χρονιά αυτή 200 εκατομμύρια έχουν ανακτηθεί από τις δημοσιονομικές αρχές. Συνήθως για να ανακτηθούν αυτά που ζητούμε εμείς που προτείνουμε χρειάζεται μια επταετία, οκταετία πολλέ φορέ. γιατί ισχύουν διαφορετικοί κανόνε. Οι δημοσιονομικέ αρχέ ξεκινούν την ανάκτηση μόνο κατά το πέρα τη δημοσιονομική χρήση. Εμεί μπορούμε τη σύσταση να την υποβάλουμε κατά την αρχή τη δημοσιονομική χρήση. Μπορεί να ξεκινάει μια πενταετία η δημοσιονομική περίοδο, αλλά η αρχή τη ανακτηση γίνεται στο τέλο τη δημοσιονομική περίοδου. Επιπλέον δεν είναι εύκολη η διαδικασία αυτή τη ανάκτηση. Μπορεί να γίνεται όχι εφάπαξ, αλλά με δόσει. Οπότε μετακυλίεται από χρόνο σε χρόνο. Δεν υπάρχει λοιπόν άμεση ε, σχέση μεταξύ των συστάσεων και της ανάκτησης. Και αν μια δεδομένη χρονιά ανακτηθούν 200 εκατομμύρια, αυτό γίνεται με βάση τις συστάσεις που έχουν γίνει πριν από μια επταετία ενδεχομένω από εμά. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ίσως περαιτέρω το σύστημα έκθεσης μας ή αναφοράς. Δεν είμαστε όμως στατιστικό γραφείο. Δεν έχουμε τέτοιους πόρους. Έχουμε περιορισμένους πόρους. Οπότε στηριζόμαστε στα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το έργο είναι τεράστιο και είναι η πρώτη φορά που ε, έχουμε τέτοια στοιχεία. Μπορούμε φυσικά να βελτιώσουμε περαιτέρω το σύστημα, ώστε να δούμε από κάθε σύσταση τι τμήμα ανακτάται τελικά και αν υπάρχει ε, υλοποίηση της σύστασης. Πάντως είναι ενδεικτικά τα στοιχεία αυτά. Τώρα, για τις περικοπές στο προσωπικό και στους πόρους γενικά, φυσικά και εμείς ε, έχουμε ε, χάσει 8 θέσεις ε, εργασίας, έχουμε υποστεί και εμείς περικοπές, έχουμε 450-500 ανθρώπους προσωπικό, υπαλλήλους προσωπικό, τα δύο τρίτα τους απασχολούνται στις έρευνες, τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο προσωπικό αφορά την πολιτική και τη διοικητικά αλλά 8 θέσεις, από όλοι 8 θέσεων είναι σημαντικός αριθμός. Οπότε 4% ε, περικοπές είναι σημαντικό ποσοστό. Έχουμε περιορισμένο προσωπικό και μεγάλο φόρτο. Γι' αυτό δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε ε, περισσότερες έρευνες. 240-250 το πολύ έρευνε ε, το χρόνο ξεκινούμε. Και η έναρξη είναι εύκολη. Η διεκπαιρέωση τη ε, έρευνα είναι δύσκολη. Δεν πρέπει μόνο να ξεκινούμε, πρέπει να ολοκληρώνουμε και τι έρευνε. Και αν το συγκρίνουμε τα στοιχεία ε, τη περσινή χρονιά πριν την αναδιοργάνωση τη ΟΛΑΦ, είχαμε 50-60% σε σχέση με το σημερινό μας έργο. Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει το τον αριθμό των ερευνών μας. Τώρα, πολιτική παρακολούθηση και συνέχιση, πολιτική συνέχεια των ερευνών, τη συνέχεια δίδεται. Κύριε Νταμάτο, ανόμεσα την ερώτηση των Πρασίνων. Τι πολιτική συνέχεια δίδεται στις συστάσεις. Εμείς δεν έχουμε πολιτικές εξουσίες, μόνο συστάσεις μπορούμε να κάνουμε και κατόπιν συντάσσουμε έκθεση για τη μη εφαρμογή των συστάσεων μας και ενημερώνουμε την εποπτική μας επιτροπή. Αλλά και η εποπτική αρχή δεν έχει αρμοδιότητες, δεν έχει εξουσίες. Αυτό προβλέπει όμως ο κανονισμός, αυτό δικαιούμαστε να κάνουμε. Εμείς, ε, επίσης, εμείς παρακολουθούμε την εφαρμογή για τις δημοσιονομικές μας τάσεις, τις ε, δικαιοδοτικές σε ό,τι αφορά τις δικαστικές συστάσεις, συνεργαζόμαστε με τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών για να διαπιστώσουμε γιατί σε μερικές χώρες εφαρμόζονται οι συστάσεις μας οι δικαστικές και σε άλλες πολύ λιγότερο. Ξεκινήσαμε με μονομένο έργο ανά χώρα για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, γιατί μπορεί εμείς να φταίμε. Μπορεί οι συστάσεις μας να μην είναι καλές ή μπορεί να φταίνουν οι χώρες να μην είναι πρόθυμες ή να μην είναι ικανές να δώσουν μια συνέχεια στις ε, δικαστικές μας αυτές τις τάσεις. Το ίδιο συνέβαινε όταν πηγαίναμε σχολείο, όταν γυρίζαμε με τον έλεγχο ε, και βλέπουμε στον έλεγχο κακούς βαθμούς, Ποιο θέλει, ο μαθητή αν έχει μόνο κακού βαθμού. Αν έχει όμω μερικού καλού βαθμού και άλλου κακού, ίσω το πρόβλημα υπάρχει και στο σχολείο. Μερικέ χώρε έχουν υψηλό βαθμό εφαρμογή των συστάσεων, άλλε χώρε πολύ χαμηλό βαθμό εφαρμογή των συστάσεων. Το συζητάμε με τους εισαγγελείς, ε, ε, με τις δικαστικές αρχές. Πάντως εμείς δεν είμαστε πολιτική αρχή, οπότε δεν μπορούμε να ασκήσουμε ιδιαίτερη πίεση. Για το οργανωμένο έγκλημα, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, μπορώ να σας δώσω μία απάντηση που είναι πολιτική βέβαια η απάντηση και σε εσάς εναπόκειται να δείτε τι θα κάνετε. Για μένα, εγώ είμαι Ιταλός βέβαια, αλλά εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχει η δυνατότητα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Ελευθεριών ε, το Κοινοβούλιο δεν έχει όμως επιτροπή που να ασχολείται με το έγκλημα. Επιτροπή Δικαιοσύνη. Εμεί έχουμε Επιτροπή Δικαιοσύνη στο Κοινοβούλιο που ασχολείται και με τι ελευθερίε και με το έγκλημα. Έτσι. Έχετε την Επιτροπή ΚΡΙΜ, εντάξει, η οποία όμως ήταν ε, προσωρινή. Έτσι δεν είναι. Καλή βέβαια μένα, αλλά περιορισμένες δια. Και κατά την ταπεινή μου άποψη, αν με ρωτάτε, και στο κοινοβούλιο τη μία πλευρά ακούμε. Ε, λοιπόν, ε, και αυτό κάτι λέει. Για την κυρία Μπρέσο, που μου έκανε ερώτηση και απαντώ αν είναι τάση, ρωτήσατε αυτή η μεγάλη αύξηση των ανακτήσεων ή αν είναι κάτι συγκυριακό. Εντάξει, η απάντηση είναι κάπου, κάπου στη μέση. Είναι αυξανόμενη η τάση μεν, αλλά όχι με αυτή την ηλικιώδη ταχύτητα όπως βλέπετε από τις 200 στις 900. Το χρόνο δεν θα είναι 900, θα είναι λιγότερο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ελαφρά αύξηση. Αν με ρωτάτε όμως, γιατί συμβαίνει αυτό, είναι περισσότερες οι απάτες, έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη ή κάτι διαφορετικό. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει αύξηση των απατών στην Ευρώπη ή στα κοινοτικά κονδύλια, ούτε καν την αύξηση, η αύξηση των ε, αιτιάσεων και των κατηγοριών. Απλώς δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και μεγαλύτερη δυνατότητα αντίδρασης και της Όλαφ και των εθνικών αρχών. Είναι πιο αποτελεσματική. Δεν σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί οι απάτες, ε, το, απλώς τις βρίσκουμε. Κύριε Βόιτσεκ, με ρώτησε κάτι. Βόλτσακ. Ε, τι διαφορά έχει η ατασταλία, η παρατυπία από την απάτη, για παράδειγμα. Αν ζητήσω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραλείπω να βάλω την ηλικία μου, γιατί επευθύνεται στους νέους το πρόγραμμα, αυτό είναι παρατυπία. Μπορεί να μην μου δώσουν τα κονδύλια είναι παρατυπία όμως αυτό. Αν πω όμως ότι είμαι 16 ετών, ενώ είμαι 45 και ξέρω πολύ καλά ότι είμαι 45 και δεν είμαι 16, αυτό είναι απάτη για να πάρω κονδύλια για τους νέους. Η διαφορά για μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί η απάτη πυροδοτεί και μια δικαστική δίωξη, διότι είναι αξιόπινη πράξη. Η παρατυπία, η ατασταλία ε, είναι λάθος, το σφάλμα ας πούμε, δεν έχει δόλο ενδεχομένως να οδηγήσει και σε ε, ας πούμε μη χρηματοδότηση προφανώς, αλλά δεν διώκεται ποινικά. Κάποιος αναφέρθηκε σε μια υπόθεση των 7 ευρώ, αυτό δεν το γνωρίζω. Εμείς δεν ερευνούμε για 7 ευρώ, ούτε μπλοκάρουμε καμία χρηματοδότηση. Συστάσεις κάνουμε για ανάκτηση. Αλλά για ανάκτηση 7 ευρώ δεν κάνουμε συστάσεις. Πώς επικοινωνούμε με τις ε, περιφέρειες. Δεν επικοινωνούμε κυρίως με περιφέρειες, αλλά με εθνικές αρχές ε, με ε, τις αρχές ε, τις δικαστικές, τις διοκτικές και τις γελικές περιφέρειες ή τοπικές αρχές ενέχονται όταν κάνουμε την κανονική μας δουλειά με την DG Regio και την DG Ample για τις αρχές που δαπανούν τα κονδύλια. Πηγαίνουμε σε κάθε χώρα για το training, την εκπαίδευση, για την ε, συνειδητοποίηση. Ε, κοιτάμε μια συνολική, μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά της απάτης και της διαφθοράς που συμπεριλαμβάνει και την πρόληψη βεβαίως, τη χρηστή ε, διακυβέρνηση, διοίκηση, δυνατότητα ανείχνευσης και αντίδρασης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ολοκληρωμένα. Κάνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη διασκέψεις, ε, εκπαιδεύσεις ε, με τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ε, με τις αρχές που δαπανούν τα χρήματα αλλά και το στοιχείο της πρόληψης. Απάντησα ασφάλματα, παρατυπίες, απάτες. Βεβαίω δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Εμείς επικεντρωνόμαστε στις κατηγορίες για πάτες. Πέντε λεπτά έχω ακόμα. Καλά, τρομερός χρόνος. Κύριε Ροπέ, για τα μεγάλα έργα, αν είναι καλύτερα επικεντρωμένα ή όχι, είναι πολιτική η ερώτησή σας, αλλά να σας απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα, σας δώσω την άποψή μου, αφού με ρωτήσατε. Από τη δική μας σκοπιά είναι καλύτερο να έχουμε απέναντι μας τις κεντρικές αρχές, γιατί είναι πιο εύκολο να επεμβαίνουμε και κανονικά, κανονικά επαναλαμβάνω, διαχειρίζονται καλύτερα τα πράγματα. Γιατί έχουν καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη οργάνωση από κάποιο δήμο ή κοινότητα. Δεν ισχύει πάντα αυτό, αλλά γενικότερα. Νομίζω είστε λετονός, έτσι δεν είναι. Τα γνωρίζετε. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη υπόθεση που ερευνήσαμε, ήταν και στις εφημερίδες. Ήταν και στη δικαιοσύνη, τη λετονική, με μεγάλη υπόθεση ενεργειακή, ε, με κοινοτικά κονδύλια, ήταν μια μεγάλη υπόθεση διαφθοράς κεντρική, τεράστια. Είναι δημόσιο, αλλά δεν θα το αναφέρω το όνομα. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν μία συνταγή. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο τοπικό είναι το επίπεδο και αποκεντρωμένο, τόσο πιο δύσκολο είναι για μας να το ελέξουμε. Αλλά την πρώτη ευθύνη για τα διαρθρωτικά ταμεία την έχουν οι κεντρικές αρχές, οι εθνικές. Έτσι εργάζεται η Ευρώπη έχουμε την αρχή της επικουρικότητας. Εάν μπορεί κάτι να αντιμετωπιστεί σε ένα τοπικό επίπεδο, αν και αν έρθει η καταγγελία σε εμά, τη στέλνουμε στις εθνικές αρχές. Δεν μπορούμε εμείς να κυνηγάμε την κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν υπάρχει κάποιος εκεί, αν δεν υπάρχει, από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς είμαστε οι αρμόδιοι δεν μπορούμε να στέλνουμε έναν υπάλληλο σε κάθε περίπτωση, αλλά για τα τα ταμεία αρμόδια είναι κυρίως τα κράτη-μέλη σε πρώτη φάση. Mr. Ε, Κυρία Μάλετιτς, τι μέτρα θα λάβουμε. Εδώ και πάλι, εμείς δεν ζητούμε περισσότερη ενημέρωση από τα κράτη-μέλη, εκτός αν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι διεθνούς χαρακτήρα ή που δεν μπορούν τα κράτη-μέλη μόνα τους να αντιμετωπίσουν. Εμείς λέμε στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζετε εσείς μόνοι σας τις περιπτώσεις, να τις διεκπεραιώνετε ε, με τρόπο αποτελεσματικό χωρίς τη βοήθειά μας και είναι και πρόθυμοι. Ε, εργαζόμαστε, ε, εκπαιδεύουμε τις αρμόδιες αρχές για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Έχουν μειωθεί οι έρευνες που ανοίγουν. Ναι, αν δείτε σε σύγκριση το 14, το 13 και το 15, τις περιπτώσεις που άνοιξαν, τις υποθέσεις, υπάρχει μείωση. μικρή όμως, 16 το αριθμό. Για μας θεωρούμε ότι είναι σταθερός ο αριθμός αυτός. Και υπάρχει αύξηση για όλα τα υπόλοιπα. Από το, έτη, από το 99. Πέρυσι είχαμε το δεύτερο ρεκόρ σε υποθέσεις. Δεν μπορούμε να κάνουν και περισσότερες, αλλά κοιτάξτε τι έγινε πέρσι. Ρεκόρ υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν στα 16 χρόνια της ζωής της Όλαφ. Στη κυρία Σμάλκοβα για την δημοσιότητα της έκθεσής μας. Εμείς, η έκθεσή μας είναι δημόσια, ε, παρουσιάζεται στα θεσμικά όργανα για πρώτη φορά και για πρώτη φορά σε αυτήν την Επιτροπή, το οποίο καλωσορίζω και ακολουθείται από συζήτηση. Όσοι θέλουν, να συζητούν. Εμείς τις θέλουν. Αλλά υπάρχουν βέβαια και συνεντευξει τύπου κτλ. Καταβάλουμε πολλές προσπάθειες για να συντάξουμε αυτές τις εκθέσει. Είμαστε λίγοι. Οι ερευνητές ε, που μετατρέπονται σε ε, ε, ειδικού τη επικοινωνία. Εγώ πιστεύω πως έχουμε βελτιώσει την ποιότητά μας. Κάθε χρόνο έχουμε πιο λεπτομερή στοιχεία, τα οποία προσπαθούμε και να εξηγήσουμε για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις. Οπότε πολλούς πόρους αφιερώνουμε εδώ και προσπάθεια και μετά οι ε, διαφερόμενοι φορείς ε, πρέπει να το χρησιμοποιήσουν και να το ξυπήσουν. Νομίζω πως απάντησα σε όλα πάνω κάτω. Είμαι στη διάθεσή σας φυσικά για άλλες συνεδριάσεις για να απαντήσω και γραπτός αν θέλετε σε επιπλέον ερωτήσεις. Και όπως είπα είμαι ανοιχτός για να έρθω για να συναντήσω οποιονδήποτε από εσά αν το θεωρείτε απαραίτητο. Ευχαριστούμε κύριε Κέσλερ. Σίγουρα είναι η πρώτη σα παρουσία και η πρώτη μα συνάντηση στην Επιτροπή Ρέτζη, αλλά σίγουρα θα είναι η τελευταία. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναπροσκαλέσουμε και να μπορέσουμε να ξαναθέσουμε ερωτήσεις. Και ευχαριστώ για την προθυμία σας να απαντήσετε και γραπτός σε κάποιες ερωτήσεις εφόσον επιθυμούν οι συνάδελφοι και γραπτέ απαντήσει στι ερωτήσει του. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Θα τα πούμε εντάχει γιατί ο χρόνο μας τελειώνει. Το τελευταίο σημείο που έχουμε προσθέσει στην ημερήσια διάταξη την κατεξοδότηση πράξη για την ενημέρωση ως προς τις ατασταλίες, την έκθεση για τις ατασταλίες. Συναφές με το έργο της Όλαφ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε ε, κατεξοδότηση πράξη δυνάμει της πέμπτης παραγράφου του άρθρου 122 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων. Η κατεξοδότηση πράξη ετοιμάστηκε από την ΟΛΑΦ ε, βάσει της βελτίωσης ε, του πρώτου τμήματος της διάταξης του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων που σας προανέφερα. Στόχος είναι ο καθορισμός των υποθέσεων ε, ατασταλιών που θα πρέπει να αναφέρονται και τι στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται με βάση το άρθρο 122.2. Έχει κοινοποιηθεί η πρόταση στο Κοινοβούλιο σε όλες τις γλώσσες 8 Ιουλίου και σας ε, στέλνει και ηλεκτρονικά σε 9 Ιουλίου. Το Κοινοβούλιο δίνεται να υποβάλει εστάσεις στην κατεξοδότηση πράξη μέσα σε δύο μήνες από την ε, ημέρα της κοινοποίηση και γι' αυτό θα πρέπει να εθετήσει το σχέδιο ψηφίσματος που, υπέβαλε η αρμόδια επιτροπή με βάση τους ε, κανόνες ε, για τις αντιρρήσεις και τις αστάσεις ε, του άρθρου 105. Και εφόσον ε, το επιθυμεί, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διμήνη παράταση. Αν ε, δεν αναλυθούν δράσει μετά την εκπνοή τη ε, προθεσμία των δύο μήνων, θεωρείται εγκεκριμένη η κατεξοδότηση πράξη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση, τη αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μα κάνει μια σύντομη παρουσίαση τη κατεξοδότηση πράξη, γιατί εμεί πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για την παράταση ή την έγκριση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για να σας παρουσιάσω αυτή την κατεξοδότηση πράξη. Και μάλιστα είναι τιμή μου να λαμβάνω το λόγο μετά την παρέμβαση του Γενικού Διευθυντού. Ονομάζομαι Μαρία Τζούνη και είμαι αναπληρώτρια τμήματάρχης της, της, της Γενικής Διεύθυνσης για την ΟΛΑΦ, ε, την ε, πρόληψη και την ανάλυση. Και το θέμα της ενημέρωσης για τις ε, ε, ατασταλίες ε, της, κα, της κάνει η ΟΛΑΦ. Γι' αυτό και η ΟΛΑΦ υπέβαλε τη σχετική κατεξοδότηση πράξη. Για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει υποχρεώσει στα κράτη-μέλη. Και μάλιστα δεν πρόκειται για μια νέα πολιτική, ο σχετικός κανονισμός που θα σας παρουσιάσω σήμερα αποτελεί τμήμα του πακέτου με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνει τέσσερις κατεξοδότηση και τέσσερις εφαρμοστικούς κανονισμούς που καλύπτουν το θέμα της διαχείρισης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Βέβαια θα ήταν καλύτερο να έχουμε μία ενιαία κατεξοδότηση πράξη, μία και μόνη, που να καλύπτει την διαχείριση, προκειμένου να έχουμε εναρμόνιση και απλούστευση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων για τις ατασταλίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη. Μια και βέβαια η ανάληψη ευθυνών, το empowerment δεν είναι ίδια σε όλες τις βασικές δράσεις, όλες τις βασικές πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τέσσερις εξουσιοδότηση κανονισμούς με τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση. Τώρα για τη συγκεκριμένη εξουσιοδότηση πράξη, όπως είπατε, αυτή καλύπτει το πρώτο τμήμα της παραγράφου 2 του άρθρου 122 του κανονισμού 1303 του 2015 που αφορά την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη-μέλη για τις ατασταλίες. Έχουμε και άλλη κατεξοδότηση δράση που αφορά την εφαρμοστέα διαδικασία για την ανάκτηση των ποσών και αυτή η δεύτερη πράξη βρίσκεται στην τελευταία φάση ε, οριστικοποίησης. Τώρα, τι ε, καινούριο έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Για πρώτη φορά έχουμε το κατόφλι της ε, υποβολής εκθέσεων της εξαίρεσης, καθώς και τον ορισμό των ατασταλιών ε, που περιλαμβάνονται στην ίδια τη βασική πράξη. Και αυτό είναι ε, σημαντικό γιατί η κατεξοδότηση πράξη γίνεται πολύ σύντομη και περιλαμβάνει μόνο τα κριτήρια της υποβολής εκθέσεων. Δηλαδή, τι ατασταλίες ε, οφείλει το κράτος μέλος να... Ε, γιατί ατασταλίες ε, οφείλει το κράτος μέλος να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε καταρχήν τις διοικητικές και τις δικαστικές έρευνες και αυτές είναι αυτές που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Και έχουμε και ένα κατάλογο πληροφοριών που οφείλουν τα κράτη-μέλη να αναφέρουν και επίσης ε, και εκθέσεις ε, παρακολούθησης, follow-up, με ειδικέ πληροφορίες συγκεκριμένε. Αυτές οι πληροφορίες τώρα, προς τι. Ε, περιλαμβάνουμε τις πληροφορίες αυτές στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσπιση των Οικονομικών Συμφερόντων. Δεν είναι έκθεση ΣΟΛΑΦ. Και εκεί γίνεται ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι αυτή η κατεξουδότηση πράξη θα πρέπει να θεωρηθεί από κοινού με την εφαρμοστική πράξη ώστε να έχουμε ισορροπημένη και ε, ε, εντύπωση και άποψη για το πακέτο των δύο δράσεων που αφορούν την υποβολή εκθέσεων και για να ε, εκπληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις από τα κράτη-μέλη για την υποβολή εκθέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών το σύστημα διαχείρισης ατασταλιών και όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει κανείς μέσω αυτού του συστήματος. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω σε απορίες. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο για περισσότερες ερωτήσεις σήμερα. Ως Πρόεδρος θα πρότεινα στα μέλη της Επιτροπής, επειδή η, εξουσιο... η κατεξοδότηση πράξη ε, διαβάστηκε πάρα πολύ αργά παραμονές ε, των θερινών διακοπών και 8 Σεπτεμβρίου λίγη η ε, προθεσμία για την ένσταση, την αντίρρηση, αν ακολουθήσουμε τους κανόνες, θα ζητήσουμε παράταση του διμήνου που προβλέπετε και θα θέσουμε την προθεσμία στις 3 Σεπτεμβρίου, 5 ώρα το απόγευμα για τα μέλη της Επιτροπής μας. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν το σχέδιο ψηφίσματος στην γραμματεία αν θέλετε να προβάλλετε αντίρρηση, η άσταση για την κατεξουδότηση πράξη και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα το διαχειριστούμε στο μέλλον. Ε, συμφωνείτε τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητούμε λοιπόν παράταση του διμήνου και το τελευταίο σημείο στη μέση διάταξη είναι οι συνεδρίες των συντονιστών σας έχουν σταλεί με email οι αποφάσεις της χθεσινής συνεδρίασης. Εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίας των συντονιστών, μάλιστα διάφορα, κανένα διάφορο. Ε, επόμενη συνεδρίαση Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί. Ευχαριστώ τους διερμηνείς εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής για τα λίγα λεπτά υπέρβασης ωραρίου. Ευχαριστώ πολύ. Λήξεις.